Colleagues, I kindly ask you... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ όσο πιο γρήγορα μπορείτε. It's already quite late, so we have to... Έχει περάσει η ώρα ήδη και πρέπει να αρχίσουμε. Thank you. Warm welcome. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε όλοι οι ευρωβουλευτές, οι σύμβουλοι, οι βοηθοί, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων, ο διερμηνής βεβαίως, λέει η κυρία Φωτίγκα. Επίσης καλώς ήρθατε όλοι μετά από την καλοκαιρινή περίοδο. Και ας αρχίσουμε τις εργασίες μας. Καθίστε πρώτα, έτσι. και όχι πηγαδάκια. Λοιπόν, αρχίζουμε την συνεδρίασή μας αυτή της μισής μέρας όπου θα εξετάσουμε διάφορα σχέδια γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων. Είναι σημαντικό το έργο μας σήμερα πάντως και πρέπει να προχωρήσουμε μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουμε. Σας υπενθυμίζω πρώτα απ' όλα ότι διαδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση αυτή, ο ήθιστε, και όσον αφορά τις γλώσσες διερμηνίας, η προτεραιότητα δίνεται στις γλώσσες των μελών που είναι πλήρη μέλη της Επιτροπής μας. Θα σας παρουσιάσω την εμερήσια διάταξη να μου πείτε κατά πόσο εγκρίνεται. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρείται εγκεκριμένη. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Θέλω να σας πω το κύριο Πάσκου, που είναι ο εισηγητής μας για την ετήσια έκθεσή μας όσον αφορά την ΚΠΑ, την Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και βρίσκεται σε ταξίδι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρόκειται για μια επίσκεψη μελέτης που κάνει στις Ηνωμένε Πολιτείες και γι' αυτό πρέπει να οργανωθούμε για να δούμε πότε θα εξετάσουμε την έκθεσή του, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό και οργανώσαμε μια επιπλέον ad hoc συνάντηση της ε, ΣΕΝΤΕ για τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου. Αυτή την ημερομηνία προτείνω τουλάχιστον. Το απόγευμα, έτσι, αργά το απόγευμα από ό,τι καταλαβαίνω. Θα δούμε πότε θα είναι. Μπορεί να είναι στις 3. 3, 3 φαίνεται ότι θα είναι. Θα σας ενημερώσουμε πάντως μέχρι τότε. Θα σας στείλουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γι' αυτό. Και τώρα περνάμε ευθύ αμέσω στο πρώτο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη και που είναι η έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας για την στρατιωτική κινητικότητα. Η συγητής μας είναι ο κύριος Τούνομ Κέλεμ από τα ΕΛΚ. Οπότε χωρίς άλλη καθυστέρηση του δίνω και το λόγο. Παρακαλώ κύριε Κέλεμ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας πω πρώτα απ' όλα ποιο είναι το πλαίσιο της έκθεσης αυτής. Είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατιωτική κινητικότητα που δημοσιεύθηκε τον Εύρεο που μας πέρασε και ακολούθησε μετά και το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο που μας πέρασε. Τώρα και τα δύο αυτά έγγραφα αναφέρονται στην τεχνική και πρακτική πτυχή της στρατιωτικής κινητικότητας. Και αυτό που λιγάκι λείπει είναι ο πολιτικός στόχος του εγχειρήματο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει προτείνει 6,5 δισεκατομμύρια μέσα και από τον προπολογισμό της διευκόλυνσης συνδέοντας για την Ευρώπη. Τα βασικά ζητήματα εδώ που αναφέρει η ανακοίνωση και το σχέδιο δράσης είναι για δίκτυα μεταφοράς και χερσαία και αεροπορικά και διαθαλάσσεις για τόσο στρατιωτική όσο και μη στρατιωτική χρήση. Υπάρχει μια ρυθμιστική χρήση τι γίνεται με τα επικίνδυνα υλικά που μεταφέρονται, τι γίνεται με τις άδειε διασυνοριακής μετακίνησης κλπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά προβλήματα, γιατί ο διάβολος βρίσκεται πάντα στη λεπτομέρεια. Το καλοκαίρι έγινε μια άσκηση με ένα όχημα χωρίς όπλα από τη Γερμανία στην Εστονία πέρασε από Πολωνία, Σλοβανία, Λετωνία και έπρεπε να συμπληρώσει ένα σωρό έγγραφα προκειμένου να προχωρήσει. Σε περίπτωση λοιπόν που βρεθούμε σε κρίση, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα σοβαρά. Γιατί παρά τις δηλώσεις που γίνονται για την αμοιβαία αρρωγή, για την αλληλεγγύη κτλ, αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα, να διασχίσουμε γρήγορα την Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση θα είναι εντελώ διαφορετική. Επίσης υπάρχει και ένα σχέδιο ΠΕΣΚΟ, μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, που σημαίνει ότι 27 χώρες, 25 χώρες μέλη αποφάσισαν να συμπεριλάβουν και την στρατιωτική κινητικότητα μέσα στα πλαίσια αυτά. Και στόχος της έκθεσής μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κυρίως να τονίσει πολιτικά το θέμα αυτό και να προωθήσει την πολιτική του διάσταση, της στρατιωτική κινητικότητας δηλαδή. Πρέπει να προωθήσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξία για να συνεισφέρουμε σε μια συλλογική αποτελεσματική άμυνα και συνεργασία από πρακτική άποψη. Πρέπει να συμπεριλάβουμε τη στρατιωτική κινητικότητα και στα διάφορα προγράμματα που λαμβάνουν χώρα εν καιρό ειρήνης. Πρέπει να αναλάβουμε δράση ώστε να μειώσουμε για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τα όποια εμπόδια και να υπάρξουν φυσικά συνέργειες και συμπληρωματικότητα με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Είναι πολύ βασικό ότι υπάρχει μια προθεσμία για να καταλήξουμε σε πολιτικές λύσεις και προτάσεις και πρέπει να τηρηθεί αυτή. Η άμυνα είναι κάτι που γίνεται σήμερα. Δεν μπορεί να καθυστερήσει και να περιμένει μεθαύριο. Και είναι και ζωτική σημασία να υπάρχει και κατάλληλη χρηματική υπηρεκοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα 6,5 δισεκατομμύρια, αν μη τι άλλο, πρέπει να παραμείνουν προκειμένου να διασφαλίσουμε την κατάλληλη μόχλευση. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις δικές σας τώρα παρατηρήσεις και σχόλια. Πρόεδρο. σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κοιόδες εισηγητές και πρώτα είναι η κυρία Ινέσα Γιάλα Σάντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σας ευχηθώ ότι καλύτερο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Και ελπίζω να μπορέσατε να ξεκουραστείτε και να είσαστε σε φόρμα τώρα και έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας μέχρι την προκλογική εκστρατεία. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον κύριο Κέλλαμ για την πρότασή του. Είναι πολύ συνολική, ενδιαφέρουσα και εγώ θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα που εκρεμεί αυτή η στρατιωτική οργάνωση. Ήταν σημαντικό ακριβώς, ήθελα και εγώ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση γιατί η μεταφορά έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί αποτελεί μία από τις αχίλιες τέρνες κατά κάποιο τρόπο ε, της Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικό το θέμα της μεταφοράς για την προστασία των συνόρων μας αλλά και για την εσωτερική μας ασφάλεια. Θα έπρεπε λοιπόν να βελτιωθεί η συνεργασία. Η στρατιωτική συνεργασία δηλαδή, που δεν είναι κάτι βέβαια καινούριο, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι είναι κάτι καινούριο. Ε, βλέπουμε ότι κάποιοι, κάποιες πλευρές δεν το θέλουν και πολύ, αλλά είναι παλιό για τις ενόπλες δυνάμεις μας. Έχουν συνεργασία στις διάφορες επιχειρήσεις τους, το βλέπουμε στους ε, δρόμους μας, αλλά υπάρχουν πράγματι δυσκολίες διασυνοριακά στις μεταφορές όπως είπε και ο εισηγητής μας. Υπάρχει καθυστέρηση. Είναι αλήθεια. Έχουμε κληρονομήσει την ιστορία μας και αυτό είναι ένα εμπόδιο. Όμως για την κοινή μας πορεία η κινητικότητα αυτή η στρατιωτική είναι πολύ σημαντική. Μόνο θετικά έχουμε να κερδίσουμε. Συμφωνώ λοιπόν ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την πρώτη προσπάθεια προκειμένου να προχωρήσει το πρόγραμμα δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα. Όλα τα στοιχεία γενικά της κινητικότητας είναι κάτι που πρέπει να έχουμε συνέχεια υπόψη μας. Τα πράγματα προχωράνε γρήγορα στις μεταφορές, η συνδεσιμότητα, οι αυτοματισμοί. Γι' αυτό και η τεχνολογία πρέπει να συμπεριληφθεί στην οργάνωση των ε, στρατιωτικών μεταφορών της στρατιωτικής κινητικότητας. Για μας είναι ζωτικής σημασίας βέβαια η πτυχή του πολίτη. Δηλαδή πάμε σε μια οικονομία κλίμακας, να μην υπάρχουν επικαλύψεις, να βοηθήσουμε να διευκολυνθεί η συνεργασία ακριβώς για να αποφεύγονται επικαλύψεις. Από την άλλη, η συνεργασία θα πρέπει να βελτιώσει γενικά την ασφάλεια και την αντίληψη που έχουμε για την ασφάλεια. Και η κινητικότητα έχει να κάνει και με τον εξοπλισμό, έτσι όχι μόνο με την οργάνωση, τη λογιστική. Υπάρχει η στρατιωτική πτυχή, υπάρχει και η μη στρατιωτική πτυχή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο πτυχών. Οι υποδομές λοιπόν, οι στρατιωτικές μπορούν να βοηθήσουν και το μη στρατιωτικό σκέλος. Πρέπει να υπάρξει επίση ενίσχυση της συντήρηση, να υπάρχει αναρμόνιση των προδιαγραφών για να χρησιμοποιούνται πιο εύκολα οι υποδομές μας, χωρίς πρόβλημα. Και μετά από αυτά που έγιναν στην Γένοβα, καταλαβαίνετε ότι οι ευθύνε μα είναι τεράστιε. Δεν πρέπει μόνο να χτίζουμε εξοπλισμό, πρέπει και να το συντηρούμε για να αντιστέκεται, για να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών. Όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Οι επενδύσεις 6,5 δις θα έπρεπε οι πολίτες να τις αντιληφθούν ότι θα πάνε όχι μόνο στους μεγάλους άξονες κινητικότητα στα διευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά ότι θα χρησιμεύσουν και σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς τους. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα ότι έτσι διασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία, οικονομία κλίμακας, συντήρηση, ασφάλεια των υποδομών και βελτίωση των προδιαγραφών στο μέλλον. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και καλύτερη οργάνωση και μείωση των εμποδίων στα σύνορα και της γραφειοκρατίας, της διασυνοριακής, υπάρχει συνεργασία του στρατιωτικού και του μη στρατιωτικού τομέα για όλες τις τεχνολογίες, αυτοματισμό κτλ. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση από την οποία όλοι θα βγούμε κερδισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Τζέφρι Βαν uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην παρούσα φάση έχω δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς στο γιατί το συζητάμε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι από το 1999 και μετά η αμυντική πτυχή της κινητικότητας και των υποδομών έχουν αποτελέσει το δικείμενο παρα... παραμέλησης τα τελευταία χρόνια. Και τώρα έχουμε βρεθεί σε μια νέα κατάσταση όπου αντιλαμβανόμαστε ότι οι αμυντικέ ανάγκες της ε, Υπήρου μα τη Ευρώπη είναι πολύ σημαντικέ. Παρακολουθείτε. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις σχετικές προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι Όλα αυτά είναι σημαντικά ώστε να μπορούμε να στείλουμε γρήγορα ε, σε επιχειρήσεις τις ε, συμμαχικές δυνάμεις σε περίπτωση σύραξης. Όλα αυτά ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία στις ε, αμυντικές μας δυνάμεις, στις δύσεις και στα αποτρεπτικά μας μέσα. Σημαντικό είναι η δυνατότητα της ενδυνάμωσης της Ευρώπης από, εξωτερικό, από το Εκτό και ε, τη Ευρωπαϊκή Υπήρου, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τι Ηνωμένε Πολιτείε και από τον Καναδά. Δηλαδή η δυνατότητα να ε, φέρουμε τις ενισχύσεις ε, εδώ και να τι κάνουμε επιχειρησιακέ. Αυτό είναι το θέμα και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Το θέμα αυτό δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, αφορά τον Νότο, τον ΝΑΤΟ ολόκληρο. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι με ποιου τρόπου θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει και πού υπάρχουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που δυσχεραίνουν το εγχείρημα αυτό και πώς μπορούμε να τα άρουμε. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ποιος είναι ο γενικότερος στόχος και ας παραμείνουμε εστιασμένοι. Σε αυτό ήθελα να επικεντρωθώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χαβιέρ Νάρτ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές, απόλυτα προφανές, ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις δεν είναι ποσοτικές, είναι ποιοτικές. Η ποιοτική τους ικανότητα ε, σημαίνει ότι μπορούν ε, να αναπτυχθούν κατάλληλα. Θωρακισμένα, μεραρχίες, πεζικό, πυροβολικό κλπ. Αν δεν μπορούν να αναπτυχθούν ε, την κατάλληλη στιγμή γρήγορα, είναι άχρηστες. Συνεπώς, αυτό που είναι βασικό είναι η ικανότητα ανάπτυξης. Αν πρέπει να υπάρξει μία επιχείρηση ή αν πρέπει να υπάρξει μία αποτροπή. Αν μπορεί να υπάρχει άμεση ικανότητα ανάπτυξης, η δυνατότητα αποτροπής είναι ζωτική σημασίας. Αν υπάρχει ένταση ή κάποιος κατακαιρματισμός που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ποτέ βέβαια με τους ανατολικούς μας ε, εταίρους, τώρα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η ικανότητα ανάπτυξη θα υπάρχει και θα είναι αποτελεσματική. Μας εξήγησε ο συνάδελφος ο αν και μένα μου ακούστηκαν κάπως ε, αλακάφκα. Δηλαδή για να γίνει ανάπτυξη δυνάμεων πρέπει κανείς λέει να περάσει από διάφορα σύνορα. Μα αυτό είναι ανέκδοτο, σαν και αυτό που λέγανε στο Χαρτούμ τότε που η Αίγυπτος πήρε το Χαλαίπ και λέγανε τότε υπάρχει πρόβλημα με την Αίγυπτο από ολόκληρο το Χαρτούμ. Μα τελικά οι Αιγύπτιοι δυσκολευόντουσαν να μπουν σε εκείνο το μικρό κομματάκι που ήταν Αίγυπτος. Ακόμα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνουμε ότι δυσκολεύεται η ανάπτυξη δυνάμων. Αυτό είναι γραφειοκρατία. Μπουροκράσια λέγεται στα ισπανικά, αλλά αν το προφέρετε διαφορετικά, μπουροκράτια σημαίνει γάιδουροκρατία, γιατί μπουρο στα ισπανικά είναι ο γάιδαρος. Έλεγα λοιπόν ότι συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Κέλλαμ. πιστεύω ότι είναι πραγματικά εξαιρετικά και το στηρίζω θα υποβάλω λίγες τροπολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν με κάτι βασικό και είναι η ικανότητα και δυνατότητα ανάπτυξης και οργάνωσης που έχει να κάνει όχι μόνο με την ευρωπαϊκή αυτονομία στο στρατό αλλά και με την ίδια τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ που αποτελεί βέβαια ένας από τους αμυντικούς μας πυλώνες. Και κάτι πολύ βασικό. Η έκθεση αυτή, παρόλο που αναφέρεται στην κινητικότητα, κινητικότητα είναι για στόχους οι οποίοι κινούνται, έτσι. Αλλά αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι οι προδιαγραφές. Γιατί αν δεν υπάρχουν κατάλληλες προδιαγραφές, υπάρχει ακινησία. Σε οποιαδήποτε επιχείρηση και ένταση, το πρόβλημα είναι η συμβατότητα των συστημάτων. Αν δεν είναι συμβατά τα συστήματα, τότε υπάρχει ακινησία. Και εδώ πολλοί δρούν εθνικιστικά και εμποδίζουν αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει λοιπόν να το εξηγήσουμε και αυτό, παρόλο που εδώ μιλάμε για κινητικότητα, ότι κινητικότητα, αν δεν υπάρχουν ενίες προδιαγραφές, σημαίνει ακινησία ή τέλος πάντων σημειωτών. Οπότε θέλω και εγώ να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία και η Ευρώπη να δείξει ότι είναι ενωμένη, όχι μόνο στο εσωτερικό της για την άμυνα υπέρ της ευρωπαϊκής επικράτειας, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει την Ευρώπη να την υποστηρίζουμε και αλλού και εκτός Ευρώπης, στο Σαχέλ για παράδειγμα, στην, ε, στο νότο της Μεσογείου, όπου εκεί στη Λιβύη για παράδειγμα υπάρχει ε, τεράστια σύγκρουση με το καθεστώς και τις διάφορες πλευρές. Λοιπόν, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να φροντίσουμε, γιατί αλλιώς θα σκάσει στα μούτρα μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν και για από τη δύναμη αυτή αποτροπής της Ευρώπης. Γιατί αλλιώ θα είμαστε ένας τεράστιος γίγαντας σε ακινησία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κλάου Μπούχνερ. Thank you very much. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Υποστηρίζουμε απόλυτα τη στρατιωτική κινητικότητα, αλλά μόνο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως περιγράφεται στο άρθρο 43 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη καλύτερες δυνατότητες ε, για μεταφορά σε περίπτωση που είναι εκτός της επικράτειας. Υποστηρίζουμε ε, την ε, αεροπορική διοίκηση στο Eindhoven που είναι μια κλασική δυνατότητα ομαδοποίησης και επιμερισμού. Λειτουργεί εξαιρετικά και δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε, να έχουμε έναν ενιαίο προϋπολογισμό στην Ευρώπη. Από αυτή την άποψη υποστηρίζουμε τον ε, εισηγητή στα όσα λέει για την ΚΕΠΑ και για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όλα τα υπόλοιπα όμως κατά την άποψή μας άπτονται των καθηκόντων των 28 κρατών μελών και του ΝΑΤΟ ε, όσον αφορά την εδαφική άμυνα. Πολιτικά και νομικά είναι πρόβλημα να ζητάμε ενωσιακά προγράμματα όπως ε, το μηχανισμό ε, τη διευκόλυνση ε, την Ευρώπη και τα 6,5 δισεκατομμύρια για μια πολιτική στρατιωτική κινητικότητα που εντάσσεται σε μια αμυντική πολιτική που αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται από τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Για να είμαι πιο ακριβή και η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή του άρθρου 42.7 τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοηθά να μιμοποιήσουμε μια τέτοια ένωση και προγράμματα ε, χρηματοδοτούμενα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Οι στόχοι της αμοιβές συνδρομής ε, δεν επιτρέπουν στην Ένωση τέτοια υλοποίηση. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και με τους σχετικούς αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΝΤΕ. Η υλοποίηση είναι καθαρά διμερής και η συνεργασία επίσης. Ε, πιστεύω ότι αυτά λοιπόν που υπάρχουν στην παράγραφο 5 είναι παραπλανητικά. Ναι, να βελτιώσουμε τις υποδομές είναι απολύτως απαραίτητο και αιτιολογημένο. Αλλά δεν βλέπουμε τι ρόλο θα έπρεπε να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Το ΝΑΤΟ και τα κράτη μέλη του θα πρέπει να κάνουν αυτό που έκαναν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Να συνεργαστούν έτσι. Αυτό είναι το βασικό καθήκον του ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουν μεταφορές, μεταφορική εταιρεία του ΝΑΤΟ. Αλλά φυσικά πρέπει να ε, απαλείψουμε όλα τα εμπόδια στις στρατιωτικές μεταφορές που υπάρχουν. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Εδώ ολοκληρώνονται οι, ε, τα σχόλια των σχεδόν εισηγητών και ανοίγουμε τη γενική συζήτηση. Mm, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω διάφορα ζητήματα. Από τη δική μου εμπειρία γνωρίζω ότι μετά από την προσχώρηση της Πολωνίας ε, το, στο ΝΑΤΟ το 1999, εγώ ανέλαβα για περίπου πέντε χρόνια την προσαρμογή των δικών μας υποδομών στα συστήματα του ΝΑΤΟ. Διαβάζοντας τώρα αυτή την έκθεση και άλλες εκθέσεις ε, προσπαθώ να τα πράγματα πρακτικά. Πέντε λοιπόν είναι τα θέματα που θα ήθελα να θέσω και τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και για τα επόμενα χρόνια, διότι πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα είναι βασικά, θεμελιώδη. Το πρώτο είναι το ερώτημα ότι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να συντονίσει τα σχέδια προσαρμογής της με το ΝΑΤΟ, με τα προγράμματα του ΝΑΤΟ. Ε, τα κράτη-μέλη, τα προγράμματα αυτά χρήση εξοπλισμών, τα κράτη-μέλη επενδύουν μεμονωμένα, αλλά υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ταμείο ε, υπό το ΝΑΤΟ στο οποίο συμβάλλουν όλα τα κράτη-μέλη και έχουν γίνει επενδύσεις μιλάμε για πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ το οποίο είναι πολυετές και πρέπει να δούμε πως το πρώτο πρόβλημα που τίθεται είναι το ότι αν εμείς θέλουμε να δαπανούμε αποτελεσματικά, να κάνουμε αποτελεσματική δαπάνη, πρέπει να δούμε το ΝΑΤΟ θα επικεντρωθεί στα δικά του προγράμματα και δαπάνες και η Ευρώπη στα δικά της. Θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος, μια μέθοδο συντονισμού για την χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην λειτουργεί ο καθένας ανεξάρτητα και χωριστά από τον άλλον. Το δεύτερο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το εξής. Αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια που προβλέπει ο επόμενο ε, προπολογισμό για την επόμενη εξαετία προβλέπουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για στρατιωτικέ απαιτήσει ή για ε, μη στρατιωτικέ και στρατιωτικέ ταυτόχρονα, διότι εδώ μιλάμε για δύο θέματα ξεχωριστά. Το να το χρηματοδοτεί μόνο τι στρατιωτικέ ε, δραστηριότητε. Εάν εμεί κάνουμε τέτοιο διαχωρισμό, προβλέψουμε τέτοιο διαχωρισμό μη στρατιωτικό και στρατιωτικό, θα μπορούσαμε ε, να ε, χρηματοδοτήσουμε και διητές ε, δραστηριότητες. Ένα τρίτο πρόβλημα. Τα κονδύλια αυτά θα χορηγηθούν για νέες επενδύσεις ή θα χρησιμοποιηθούν και για τον εξυγχρονισμό ήδη υπάρχουσων υποδομών. Όσον αφορά τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα και την εξοικονόμηση χρημάτων, καλό θα ήταν να προβλέψουμε και την αναβάθμιση ε, και την ανακαίνιση παλαιών υποδομών. Μην το ξεχνάμε αυτό το ερώτημα. Μετά, οι διασυνοριακές επενδύσεις. Διότι έχουμε σύνορα που αποτελούν εμπόδια όχι μόνο νομικά αλλά και τεχνικά. Ήθελα λοιπόν να μάθω κατά πόσο ενδεχομένως τα διαθέσιμα κονδύλια θα μπορούσαν ενδεχομένως να επικεντρωθούν στις διασυνοριακές επενδύσεις. Γιατί το λέω αυτό. Διότι ήδη έχουμε κάποιες προτάσεις ε, τροποποίησης της χρήσης αυτών των 6,5 δισεκατομμυρίων. Εάν ε, δεν εγκρίνουμε αυτή τη χρηματοδότηση θα δώσουμε ε, την εντύπωση ότι αυτή είναι η χιλιοστή επένδυση σε υποδομές. Ε, δεν θα χρησιμοποιηθεί επαρκώς αυτό το κονδύλιο, αυτό το Ταμείο Χρηματοδότησης για τις ενεργητικές απαιτήσει. Ένα άλλο πρόβλημα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, βασικός χρηματοδότης είναι η Ευρωπαϊκή Τραπεζά Επενδύσεων, η οποία διαθέτει τεράστια κονδύλια τα οποία ε, συμπληρώνουν ε, τις ε, επενδύσεις σε υποδομές. Και το πρόβλημα είναι ότι το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν μπορεί να χρηματοδοτεί στρατιωτικές δραστηριότητες. Αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και απαιτεί κάποια άμεση δράση και κάποια συζήτηση για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Σας ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή. Και ακούγοντά σα, αναρωτιέμαι ποια μέθοδο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε στο μέλλον ε, για να υπερβούμε όλα αυτά τα προβλήματα, για να δώσουμε απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Σίγουρα θα το συζητήσουμε και με την γραμματεία και με του συντηρηστέ για να δούμε κατά πόσο είναι δυνατό να γίνει μια συζήτηση με τους αρμόδιους συναδέλφους ε, στα τμήματα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο ΝΑΤΟ. Ίσως θα τα καταφέρουμε και φέτος, εντός του έτους. Ευχαριστώ. Outmans. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή πρωτοβουλία, η οποία έρχεται μια πολύ καλή στιγμή. Θα ξαναμιλήσουμε βέβαια για την στρατιωτική κινητικότητα αργότερα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια καλή έκθεση. Τονίζει ότι η στρατιωτική κινητικότητα τη σήμερον ημέρα είναι ζωτική σημασία την εποχή αυτή που ζούμε Άρα πρέπει να διευκολύνεται. Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι οι εναρμονισμένες προδιαγραφές. Αυτό πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Εάν θέλουμε η Ευρώπη να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί και η κινητικότητα αυτή να λαμβάνει χώρα γρήγορα, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και μαζί να φροντίσουμε να μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η στετιωτική κινητικότητα χωρίς εμπόδια. Βέβαια, οι χώρες μέλη μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και η Ευρώπη έχει να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε, με τον συνάδελφο Όναρτ συμφωνώ επίσης ότι η έκθεση έρχεται σε μια πολύ καλή στιγμή και ότι πρέπει να συνεργαστούμε ότι στην πράξη γρήγορα να τεθούν σε εφαρμογή όσα αναφέρει η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Φρόντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κέλαμ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπω σε λεπτομέρειες. Θα περιοριστώ μόνο στο ότι είναι εκπληκτικό αυτό που μαθαίνουμε, ότι δηλαδή τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ μπορούν να κινηθούν στην ε, επικράτεια της ε, Ευρώπης ανεμπόδιστα. Ενώ παράλληλα τα ευρωπαϊκά στρατεύματα, όπως μας εξηγήσατε, πρέπει να συμπληρώσουν πέντε διαφορετικά έγγραφα για να περάσουν σύνορα και να πληρώσουν και φόρους μάλιστα. Αν καταλαβαίνω καλά αυτό το σύστημα. Όμως, θα κάνω μια πολιτικού χαρακτήρα παρατήρηση, μια ευρύτερη παρατήρηση. Ο κύριος Βαν είπε, και δυστυχώς λείπει τώρα, ε, ότι Εμείς δεν θέλουμε να εξηγήσουμε την κάθε μας πράξη, αν κατάλαβα καλά. Και στόχος είναι να δημιουργήσουμε μία αξιόπιστη ευρωπαϊκή στρατιωτική άμυνα. Αλλά δεν ξέρουμε τι προκάλεσε αυτές τις ε, νέες εξελίξεις, ούτε αναφέρθηκε το όνομα του Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος πάνω από μία φορά άφησε να εννοηθεί ότι μέσα σε μια στιγμή μπορεί να αποσύρει όλα τα στρατεύματα των ΗΠΑ από την Ευρώπη. Και επίσης μην ξεχνάμε και τις εξελίξεις στα ανατολικά μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς και να αρνούμαστε το ότι η Ρωσία έχει εισβάλει στην Κρυμαία, η Ρωσία εμπλέκεται στην Ανατολική Ουκρανία και όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτω σχέση με την επανεξέταση του αμυντικού συστήματος στην Ευρώπη. Δεν ξέρω λοιπόν ε, αν θα ήταν κατάλληλη στιγμή να εκφράσουμε με σαφήνεια τους στόχους μας. Είτε αυτό είναι καλό, είτε αυτό όχι. Αυτό βέβαια είναι στην κρίση των μελών της Επιτροπής. Θεωρώ όμως ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να μην ε, κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας και να μιλάμε με ξεκάθαρο τρόπο. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, ο κύριος Ντρογεύσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοι, να επανέλθω όμως και σε αυτά που είπε ο κύριος Νάρτ. Θεωρώ πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η συμβατότητα, η τυποποίηση και η επάρκεια. Αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος για όλα αυτά στις ε, δυνάμεις του ΝΑΤΟ και σε εκείνε των κρατών μελών της Ένωσης. Θεωρώ όμω ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο, διότι παρατήρησα διάφορα προβλήματα διοικητική μέρημνα ε, στη μεταφορά εξοπλισμού, ε, πεζικού, ιατρικών προμηθειών κτλ. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα ε, όχι έλλειψης συμβατότητας ανάμεσα στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μη συμβατότητα με τις τρίτες χώρες. Και μην ξεχνάμε πως ε, δραστηριοποιούμαστε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάμαι μάλιστα, κατά την πολιορκία του Σαράγεβο, η Ουκρανία είχε δώσει αεροπλάνα για να μεταφερθούν ιατρικές προμήθειες μεταξύ άλλων. Και τα αεροσκάφη αυτά δεν ήταν συμβατά με τα συστήματά μας. Και πολλές φορές έπρεπε να αυτοσχεδιάσουμε για να εξαναγκάσουμε ε, αυτά τα σκάφη να γίνουν συμβατά. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν ε, όχι μόνο τα νομικά ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα συμβατότητας, επάρκειας και τυποποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο ξανά στον κύριο Κέλαμ, τον εισηγητή, για τα καταληκτικά του σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Εκτιμώ πολύ τα θετικά σας σχόλια και τη θετική σας στάση Ελπίζω λοιπόν η έκθεση να γίνει ακόμα καλύτερη χάρη στη συνεισφορά σας. Το κυριότερο που έχει προκύψει από την συζήτηση αυτή είναι το θέμα της κινητικότητας. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα στην πράξη. Η στρατιωτική κινητικότητα δεν αντιτίθεται στις ε, ανάγκες ε, των ε, πολιτών και για να την βελτιώσουμε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν θα εξυπηρετεί μόνο στρατιωτικούς αλλά και πολιτικούς σκοπούς. Δεν είναι αντίθετες αυτές οι έννοιες. Εσείς κύριε συνάδελφε, μας δώσατε ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι σημαίνουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην περίπτωση της Αιγύπτου. Πολλές φορές η γραφειοκρατία, ξέρετε, είναι το καλύτερο όπλο εναντίον του αντιπάλου. Και είναι πολύ κέριο αυτό που είπατε. Στόχος είναι η ανάπτυξη δυνάμεων την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο μέρος. Το θέμα βέβαια είναι πώς θα το επιτύχουμε στην πράξη. Ε, ο κύριος Βανόρντεν επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη κατανόησης ε, της ε, βοήθειας που φτάνει στην Ευρώπη από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αυτό όμως που δεν ήταν σαφές είναι η υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 6,5 δις θα καλύψουν μόνο τη στρατιωτική κινητικότητα ή και πολιτικές ανάγκες. Αυτό δεν ήταν σαφές. διότι η επιθυμία όλων είναι να μην διατεθούν αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια μόνο σε στρατιωτικές ανάγκες. Και μία άλλη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει τέτοια έργα. Νομίζω πως ε, αυτά είναι εύλογα ερωτήματα και όπως είπατε κι εσείς μπορεί να μην είναι δυνατόν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, όμως πρέπει να το δούμε. Ε, κύριε Φρόιντ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με το ότι πρέπει να τονίσουμε ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης ευρωπαϊκής άμυνας και ότι αυτό δεν αντιτίθεται στους στόχους του ΝΑΤΟ. Αλλά όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν με τις ΗΠΑ, για παράδειγμα, θα έπρεπε να προκαλέσουν θετικές αντιδράσεις από τη δική μας μεριά, έτσι ώστε εμείς να φροντίσουμε τη δική μας άμυνα. Και φυσικά δεν είναι προνομιούχο το ΝΑΤΟ, χρειάζεται να ε, συμμορφώνεται στις ίδιες απαιτήσει με ε, τις δυνάμεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι αντιμετωπίζουν, θεωρώ, την ίδια γραφειοκρατία. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Ε, θα χαρώ να λάβω τροπολογίες και προτάσεις έτσι ώστε να ε, βελτιώσουμε την έκθεση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 12η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Σε μια εβδομάδα περίπου δηλαδή. Έχετε μια εβδομάδα καιρό για τροπολογίες. Δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο στην ε, συνεδρία της Επιτροπής μας στις 10 ή 11 νομίζω του μηνός. Στην άφετη έκθεση θα εγκριθεί στις 5 Νοεμβρίου και λογικά στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για το σημείο αυτό. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή της έκθεσης για την, ε, της έκθεση για τη λειτουργική διάταξη σχετικά με τις εξαγωγές όπλων. Κυρία Λόζινγκ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να ξεκινήσω λέγοντας ότι η παρουσίαση της έκθεσης μου σχετικά με την κατάσταση της ε, υλοποίησης της κοινή ε, θέσης δεν έχει αλλάξει και πολύ. Και αυτό συνεπάγεται ότι δεν έχουν αλλάξει και πολύ οι προτάσεις για βελτίωση της κοινή θέσης. Όμως, αυτό το νομικά δεσμευτικό όργανο έχει ακριβώς αυτόν τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τα προβλήματα είναι πολλά σχετικά με τις εθνικές εξαγωγές όπλων και διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Οι διαφορές επίσης βρίσκονται και στην ερμηνεία ε, του κειμένου, του νομικού κειμένου. Οι εξαγωγές όπλων έχουν, συνεχίζουν να έχουν ελλειπή δεδομένα. Τα ελλειπή δεδομένα οφείλονται εν μέρη και στην ε, ασάφεια ως προς την ερμηνεία του κειμένου. Όταν δεν υπάρχουν ενιαίες ε, και όταν οι εκθέσεις που παίρνουμε από τα κράτη-μέλη διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, αυτό ε, βλέπουμε ότι δημιουργεί πρόβλημα και όσο δεν υπάρχουν συνέπειες, ε, τα προβλήματα εντείνονται. Επίσης, θεωρώ λυπηρό ότι στην παρούσια έκθεση δυστυχώς αναφέρονται τα στοιχεία για τις εξαγωγές όπλων το 2015 και το 2016. Δεν έχει γίνει καμία ε, ποιοτική ανάλυση των δεδομένων από την στιγμή που αυτά συλλέχθηκαν και δημοσιεύθηκαν. Για τους λόγους αυτούς, επαναλαμβάνουμε την ε, αίτηση της ε, κυρίας Βαλέρο που συνέταξε την προηγούμενη έκθεση για βελτίωση της διαδικασίας ε, συλλογής και διαβίβασης των δεδομένων. Το αργότερο τον Ιανουάριο του ε, επόμενου έτους ε, από τη συλλογή των δεδομένων. Αυτά θα πρέπει να δημοσιεύονται. Πρέπει να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες προθεσμίες. Ε, το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο θα πρέπει να έχουμε τα δεδομένα δημοσιευμένα. Μετά, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων για το 2016 και το 2017. Το 2013 έως το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε εξαγωγές όπλων που ανέρχονταν στο 27% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι μυστικό. Ο στόχος βέβαια των εξαγωγών ε, ήταν περιοχές ε, στις οποίες ε, υπάρχουν συγκρούσεις, περιοχές που βρίσκονται σε κρίση. το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών αυτών πήγαινε στις, ε, στη Σαουδική Αραβία και στις χώρες της με, Μέσης ε, Ανατολής. Και το 57,9 57, δις κατέβαλαν ε, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για εισαγωγές όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατιωτική τεχνολογία που εξάγεται λοιπόν σε αυτά τα ε, κράτη χρησιμοποιείται για σκοπούς που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας και των εξαγωγών αξίζει να σημειωθεί ότι το 95% των ετήσεων ε, εξαγωγών ε, όπλων ML9, πολεμικά σκάφη δηλαδή, εγκρίθηκαν. Τα σκάφη αυτά χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό της Ιεμένης. Και αυτός ο θαλάσσιος αποκλεισμός έχει οδηγήσει ε, στο θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων, σε άλλους τόσους να ζουν σε άθλιες συνθήκες. Και αυτός ο εξοπλισμός έχει ε, φτάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται επομένως μεγαλύτερος έλεγχος, μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτά είναι απαραίτητα. Και ε, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της κοινή μας ε, θέσης ε, θα πρέπει να χρησιμοποιείται γλώσσα ξεκάθαρη, σαφέστατη έτσι ώστε να αποφευχθούν οι διαφορετικές ερμηνείες των κριτηρίων. Ο τομέας της άμυνας και η Αμυντική Ένωση είναι πολύ ε, βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μάλιστα με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας αυτό κατέστη ακόμα σαφέστερο. Και στο πλαίσιο όλων αυτών θα πρέπει να επανεξετάσουμε την χρηματοδότηση των έργων που ε, θα χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και, και στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής Ασφάλεια και άμυνας και θα πρέπει να διασφαλίζεται ο ε, απόλυτος ε, έλεγχος. Ακόμα και το μέσο της, ε, για την ειρήνη, το οποίο ανακοίνωσε ε, η Επίτροπος ε, Μογκερίνη με, που θα προβλέπει εξαγωγές ε, εξοπλισμού στις ε, συμμαχικές μας χώρες. Αυτό πρέπει να το επανεξετάσουμε. Αυτά προς το παρόν από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος του Νομικέλεμ είναι ο πρώτος και εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την έκθεση αυτή, η οποία, όπως ξέρουμε, δεν ε, υποστηρίζεται ομόφωνα. Υπάρχουν κάποιες αρνητικές πτυχές. Νομίζω ότι η έκθεση τονίζει ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη από δύο πλευρές. Λέει ότι δεν εφαρμόζουν τα κριτήρια της κοινή θέση, δεν υπάρχουν μηχανισμοί κυρώσεων και από την άλλη μεριά δεν παρουσιάζουν έγκαιρα τις ε, αναφορές τους. Τώρα είναι θέμα προσέγγισης. Πρέπει όντως να name and shame, να καταδεικνύουμε δηλαδή και να δακτυλοδεικτούμε ποιος φταίει ή πρέπει να ακολουθήσουμε μια πιο ήπια προσέγγιση. Η έκθεση κατά κάποιο τρόπο Αναρωτιέται για τα άρθρα 7 και 8 και το 9 που λέει ή για τη μεταφορά των προϊόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένει ότι οι μεταφορές αυτές πρέπει να είναι συνεπείς με την κοινή θέση. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε πολύ στα σοβαρά τα προβλήματα ε, του ελέγχου όπλων, κυρίως των όπλων που είναι παράνομα και ξεφεύγουν του ελέγχου μας. Από την άλλη πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για τη συλλογική ε, αμυντική ικανότητα της Ευρώπης. Την ανάγκη για ανανέωση. Συνεπώς το ΕΛΚ θα υποβάλει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση για τα κράτη-μέλη κυρίως. Και υπενθυμίζω ότι η κοινή θέση είναι μια δήλωση που, με την οποία παραμένει η αρμοδιότητα στις χώρες μέλη. Ού μας πάτε τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια για την παρουσίασή της. Κατά τη γνώμη μας η έκθεση αντιμετωπίζει προβλήματα που είναι παρόντα στον κόσμο μας και λαμβάνει υπόψη τις γεωπολιτικές αλλαγές βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι περισσότερο παρούσα στην αμυντική πολιτική. Είναι σαφές ότι πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλειά μας όλο και περισσότερο στην Ευρώπη. Οπότε μας εκπλήσει ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό αδειών εξαγωγών από τότε που αρχίσαμε να συλλέγουμε στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δείχνει ότι τελικά οι χώρε μέλη δεν ακολουθούν την κοινή θέση. Υπάρχει πρόβλημα επίσης με τις χώρες μέλη, οι οποίες δεν αναφέρουν ε, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν τα στοιχεία τους. Βλέπουμε ότι αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα, από εκεί που έχουμε στοιχεία δεν τηρούνται παντού τα αυτοκριτήρια. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το 7,2% των αιτήσεων αδειών για, έξω, για εξαγωγές στην Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για παράδειγμα εγκρίνονται ενώ οι χώρες αυτές παραβιάζουν έξω από τα αυτοκριτήριο της κοινή θέση. Θα πρέπει να τους αρνούμαστε τις ε, εξαγωγές αυτές. Αλλά δεν υπάρχει μηχανισμός κυρώσεων Οπότε χρειαζόμαστε κοινή ερμηνεία των οχτώ κριτηρίων, χρειαζόμαστε ένα κοινό σύστημα αναφοράς και χρειαζόμαστε και κυρώσεις σε βάρος όσων δεν ακολουθούν την κοινή θέση. Έπειτα, οι τρεις χώρες, μερικές έχουν αποφασίσει να ακολουθούν την κοινή αυτή θέση και πρέπει να τις στηρίξουμε αυτές κατά προτεραιότητα στο δρόμο τους προς την Ευρώπη, εφόσον τηρούν την κοινή αυτή θέση για τις εξαγωγές όπλων. Έπειτα τα θέματα ε, που αποτελούν μεγάλη πρόκληση για μας είναι και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να διαθέσει αρκετά κονδύλια και ανθρώπινο δυναμικό και να εκπαιδεύσει προσωπικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ μας προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ήταν η τελευταία παρέμβαση σχεδόν εισηγητών. Τώρα η γενική συζήτηση, κύριος Αρνελίτς πρώτος. δεν μα είχε κοινοποιηθεί, συγγνώμη. Αλλά έτσι κι αλλιώ είδατε, δεν έκλεισα τη συζήτηση, συνεχίζεται έτσι. Η κυρία Βαλέρο είναι στη Σουηδία που είναι η σκιώδη συζήτητριά μα και την αντικαθιστώ. Αλλά θα είμαι πολύ σύντομο. Καταρχά κυρία Λόζινγκ, θέλω ήθελα να σα συγχαρώ ε, θερμότατα για την ε, πολύ καλή έκθεση. Καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή, όλα όσα λέγονται στην έκθεση αυτή. Πάντα βέβαια, μας ξέρετε, η κυρία Βαλέρο πάντα έχει να προσθέσει κάτι. Και εδώ φαντάζομαι θα κάνει το ίδιο. Εγώ θα σταματήσω και ξέρετε και από την προηγούμενη φορά τι θα ήθελε και εδώ να προσθέσει. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε. Ο κύριος Αρνελίτς τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε εγώ είμαι σκιώδης για τους σοσιαλιστές, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Λουζίν για αυτή την ισορροπημένη έκθεσή της. Συμφωνώ με τα περισσότερα πράγματα που λέτε, κυρίως για το ότι πρέπει να υπάρχει ένα σώμα που να φροντίσει για την συνεπή εφαρμογή και τήρηση της κοινή θέση. Να υπάρχει και κοινοβουλευτικό έλεγχο για τι αποφάσει όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών. Πρέπει να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί δίνουμε τα χρήματα, αλλά δεν ελέγχουμε. Μα πρέπει και να μπορούμε να ελέγξουμε. Γενικά, κάνω έκκληση για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώ ελέγχου των εξαγωγών. Αν δεν υπάρχει αυτό δεν μπορούμε να έχουμε καν κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Έχουμε να κάνουμε με μια νέα απειλή, μια νέα κατάσταση. Έχουμε την Ρωσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσει τόσο συμβαίνουν σήμερα και να σας υπενθυμίσω ότι ευρωπαϊκά όπλα δόθηκαν και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές στη Συρία. Είναι ένα παράδειγμα το που καταλήγει η εξαγωγή όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό χρειάζεται συνοχή και δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να ζητήσουμε και να το τηρήσουν οι χώρες μέλη. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για τη διπλή χρήση και να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Η έκθεση είναι καλή. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια δεν μπορούν πλέον να εξαχθούν. Αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παλιά αποτελούσαν ένα εμπορεύσιμο αγαθό. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την επιτυχία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό να επιμείνουμε περισσότερο και όσον αφορά τις εξαγωγές ε, όπλων. Θα υποβάλουμε διάφορες ε, τροπολογίες και προσβλέπουμε και εμείς τη συζήτηση που θα γίνει στο Κοινοβούλιο. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η κυρία Λέζινγκ και πάλι για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την πλειοψηφία των ε, σχολείων. Γι' αυτό θα περιμένω με χαρά τις ε, τροπολογίες που θα βελτιώσουν την έκθεση. Ε, κύριε Κέλλαμ, θα ήθελα να σχολιάσω ότι η ομοφωνία που αναφέρεται. Ή έλλειψη μάλλον αυτοίς στην παρατήρησή σας έχει ως αφετηρία την έκθεση της κυρίας Βαλέρο, η έλλειψη μάλλον αυτής στην παρατήρησή σας έχει ως ε, αφετηρία την έκθεση της κυρίας Βαλέρο, η οποία εγκρίθηκε με πλειοψηφία. Και δεν έχει αλλάξει η βασική προσέγγιση της έκθεσης ε, από την προηγούμενη συγκήτρια σε μένα ο προσανατολισμός ε, δεν είναι σαφέστατα εναντίον της αμυντικής βιομηχανίας. Η έκθεση απαιτεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και τα σημεία τα οποία αναφέραμε ε, είναι στοιχεία, γεγονότα και όχι ε, κατονομάζουμε, δακτυλοδεικτούμε ορισμένους. Αυτό όσο προς το σχολείο σας και προσβλέπω στην συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται το σημείο αυτό. Σας ενημερώνω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Στις 12 το μεσημέρι. Έγκριση στην ΑΦΕΤ αρχές Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου. και ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι η πρώτη εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Η συγητής είναι ο κύριος David Μακάλιστερ. Εδώ θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε το ονόματα των σχεδόν που υπέδειξαν οι πολιτικές ομάδες. Οι πολιτικές ομάδες, από όσο γνωρίζω, καθυστέρησαν λίγο στην υποβολή των ονομάτων των σκιωδών. Υπήρξαν λοιπόν κάποια προβλήματα με αυτό. Χωρίς άλλη καθυστέρηση ας ξεκινήσουμε. Κύριε Μακάλιστερ, παρακαλούμε. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησης σε πρώτη εξέταση. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω το σχέδιο γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας εδώ στη ΣΕΝΤΕ. Όπως γνωρίζετε, η ΙΤΡΕ είναι η επί της ουσίας ε, ε, ε, επιτροπή, ο κύριος Κρασνοτεύσκη Εμεί είμαστε συνδεδεμένοι Συνδεδεμένη Επιτροπή τη διαδικασία του άρθρου 54 όπω επεσήμανε η πρόεδρο το ημερολόγιο με την Ήτρα έχει συντονιστεί ω εξή. προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 13η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι είναι μικρή η προθεσμία αλλά όπως θα δείτε είναι αναγκαίο για να μην καθυστερήσει όλη η διαδικασία εξέταση των τροπολογιών στη συνεδρίαση της ΕΝΤΕ στις 10 Οκτωβρίου ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα λάβει χώρα στις 5 Νοεμβρίου. Η Ήτρα θα ψηφίσει τη γνωμοδότηση στην 21η Νοεμβρίου και η εντολή για τον τριμερή διάλογο θα ψηφιστεί στην Ολομερία του Δεκεμβρίου ώστε να, ξεκινήσει, να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι ε, το 2019 για τη γνωμοδότηση Έχω κάνει κάποιε προτάσει για την προτινόμενη ηθική εξέταση των προτάσεων Κομισιόν. Ούτε έχει δώσει ορισμό, ούτε έχει σχεδιάσει επαρκώ την εξέταση. Ελπίζω ότι η πρότασή μου θα μπορέσει να συμβάλλει θετικά στη συζήτηση. Η ουσία πρέπει να είναι ότι η Κομισιόν θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι προτάσεις υποβάλλονται συστηματικά σε εξέταση διοντολογίας ηθική εξέταση ώστε να έχουμε ισότιμες ε, συνθήκες ανταγωνισμού αφού όλα αυτά συζητηθούν και η συμφωνία ε, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Ε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε στη συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για να επιτύχουμε κάποιες πλειοψηφίες. Επίσης θέλω να ενισχύσουμε τις αναφορές στις δυνατο... δυνατότητε. στο σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η στρατιωτική αυτονομία δεν, δεν αναφέρεται μόνο στην έρευνα αλλά και στις επιχειρήσεις. Εδώ η πρόταση της Κομισιόν είναι κάπως ε, ασαφής. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς εννοεί με την αμυντική βιομηχανία και την άμυνα. Θέλω να είμαι βέβαιος ότι ο κανονισμός θα καλύπτει και τα δύο επαρκώς τρίτων Κάτι που με ανησυχεί είναι το ζήτημα των τρίτων χωρών. Αυτό περιλαμβάνει διάφορε διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αφορά χώρες που θέλουμε να είναι μέσα. Προς το παρόν έχουμε την Νορβηγία. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέσα ή ίσως όχι. Ανάλογα με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Brexit, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει λόγος να συμπεριλάβουμε κάποιο ρήτρα για το Ηνωμένο Βασίλειο δίπλα στην Νορβηγία. Ε, πρέπει να συζητήσουμε την εμπλοκή του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα που θα πρέπει να συζητηθούν εκτενώς. Η δεύτερη διάσταση αφορά το επίπεδο ελέγχου που μπορεί να έχουν τρίτες χώρες ε, στα δικά μας προγράμματα. Αυτό που με ανησυχεί εδώ είναι ότι μπορεί να μην έχουμε αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα. Το ζήτημα των αδειών εξαγωγών τρίτων χωρών όπως ο κανονισμός για το διεθνές εμπόριο όπλο των ΗΠΑ που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την έκβαση των προγραμμάτων μας στο μέλλον εάν δεν το αντιμετωπίσουμε επαρκώς. Εγώ έχω προτείνει κάποια πράγματα για να λύσουμε αυτό το θέμα. Τέταρτον, η αδειοδότηση εξαγωγών εντός της Ένωσης είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Για τους σκοπούς του προγράμματος αυτού προτείνω να χρησιμοποιήσουμε το Γενικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων Μεταφορών από τη σχετική οδηγία. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία αυτή εδώ και χρόνια, κάτι που θα μειώσει σημαντικά τον ε, γραφειοκρατικό φόρτο ε, το να χρησιμοποιηθούν αυτές οι άδειε μεταφοράς. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε κράτος μέλος θα δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα του μια γενική άδεια συνεργασίας με επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση κατά την ανάπτυξη προτάσεων έργου στο πλαίσιο του EDF. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ενημερώνουν τις σχετικές ε, αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, χωρίς όμως να χρειάζεται να ζητήσουν προηγούμενη άδεια. Και τα κρατημέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν άδειε όταν να πλήττονται τα συμφέροντά τους. Και πέμπτον, καταλαβαίνω ότι ορισμένοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη συμφωνήσει ε, για το EDIDP και για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ε, για θέματα επιλεξιμότητας. Δεν έχω κάνει προτάσεις γι' αυτό, αλλά ευχαριστούμε να το εξετάσουμε. Μία τελευταία παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε. Μου είπαν ότι γίνονται αυτή τη στιγμή συζητήσει μεταξύ νομικών εμπρογνωμόνων στο Κομισιόν και στο Συμβούλιο για να χωρίσουν το ενίο Ταμείο Άμυνα από τον Ορίζοντα Ευρώπη. Θέλω να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μας ε, δημιουργήσει πρόβλημα στις συζητήσεις. Συγγνώμη που μακρηγόρησα την επόμενη φορά που θα πάρετε το λόγο εσείς ε, ε, να μιλήσετε περισσότερο. Κανένα πρόβλημα εκ μέρους των σοσιαλιστών ο κύριος Τονινού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πάσκου, που είναι σκιώδης ηγητής ε, των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, λείπει, οπότε θα παρουσιάσω εγώ τα σχόλιά του για την γνωμοδότηση αυτή. Ε, χαιρετίζουμε λοιπόν την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνα στο επομενο πολιτες πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. ακολουθεί τον κανονισμό EDIDP και στόχο έχει να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που θα διασφαλίσει συνέχεια χρησιμοποιώντας ήδη ένα μέρος ε, από το κείμενο του κανονισμού EDIDP που το που δημοσιεύτηκε το πρώτο εξάμεινο του 2018. Ωστόσο, η διαφορά είναι σημαντική με την έννοια ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ε, αποτελεί ε, ένα μέσο στο πλαίσιο του οποίου θα δημιουργηθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Θα ασχολείται με ε, δύο τομείς ε, έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων. Καταρχάς, έχει έναν αρκετά γεννόδωρο προϋπολογισμό. 13 δισεκατομμύρια έχουν προταθεί και 4,1 δισεκατομμύρια για την ε, αμυντική έρευνα, 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ για ανάπτυξη ικανοτήτων. Έπειτα, θα υπάρχει συνέργεια με άλλα προγράμματα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και θα υπάρχει και μια συμπληρωματική εργαλειοθήκη που στόχο θα έχει ε, απόκτηση αμυντικής τεχνολογίας και αμυντικών προϊόντων από τα κράτη-μέλη ως αποτέλεσμα των ε, προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Ε, το σχέδιο γνωμοδότησης ε, που συνέταξε ο κύριος Μακάλιστερ συνεχίζει την ε, πρόταση αυτή και την πηγαίνει ακόμα παραπέρα. Ασχολείται με, το θέμα των, της χορήγησης αδειών, ε, της αμυντικής έρευνας για προϊόντα και τεχνολογία ε, δημοσιονομικές συνέργειες με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ε, πτυχές στρατιωτικής εκκινητικότητας στα πλαίσια του Connecting Europe. Στόχο έχει να ε, παρακολουθεί τις αναδυόμενες νέες τεχνολογίες και να υπάρχει, να αλληλοσυμπληρώνονται τα διάφορα ταμεία. Ωστόσο, θα υποβάλουμε τροπολογίε την επόμενη εβδομάδα και θα σας αναφέρω μόνο δύο από αυτές. Πρώτον, χρειάζεται καλύτερη αναφορά στις διατάξεις του κανονισμού EDIDF ε, για την ε, συνεργασία με άλλους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ. Και έπειτα θα θέλαμε να αποφύγουμε την διάταξη που απαιτεί τουλάχιστον τρία, ε, τρεις οντότητες από τρία κράτη-μέλη ε, να συνεργάζονται για να ληφθεί χρηματοδότηση ε, από το Ταμείο. Στόχος του κανονισμού EDIDP είναι να ενισχύσει την ε, διασυνορική και διεθνή συνεργασία στα αμυντικά ζητήματα. Και ε, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι με τον κύριο Μακάλιστερ ε, θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να καταρτήσουμε ε, μια ως το δυνατόν καλύτερη γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΑΦΕΤ και τον κανονισμό DIDP. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Να κάνω μια ερώτηση. η Ο κύριος Πράιτ από τους φιλελεύθερους ήταν σκιοδησηγητής. Όχι, δεν είναι εδώ. Ωραία, η κυρία Λόζιν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εστιάσω σε μια συγκεκριμένη πτυχή. Αυτή τη στιγμή η η γνωμοδότησή μας ε, έχει σχέση και με μία έκθεση που συζητιέται στην Επιτροπή Ήτρε. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να συμφωνήσω και με τον κύριο Μακαλίστερ και με την κυρία Φωτίγκα. Αυτό το ταμείο θα ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι μια πολύ, ένα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο των εκθέσεων και της Επιτροπής ΑΦΕΤ και της Επιτροπής ΙΤΡΕ. Και να σας Υπενθυμίσω την επιστολή της ε, Πρόεδρου Φωτίκα και του κύριου Μακάλιστερ στην, Επίτροπο Βίξτρομ από το, ε, στην Πρόεδρο Βίξτρομ από το 2017, η οποία αναφέρει ότι το άρθρο 52 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στην, ε, στην στρατιωτική συνεργασία και την πολιτική συνεργασία για αμυντικά ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν αρκετά λυπηρό το ότι αυτό ε, δεν ελήφθη καθόλου υπόψη το άρθρο 52, διότι εδώ Υπάρχει παραβίαση του άρθρου 41.2, το οποίο απαγορεύει ε, χρηματοδότηση από τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στρατιωτικών προγραμμάτων που στόχο έχουν την επίθεση σε άλλες χώρες ή την στήριξη συγκρούσεων. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να τηρούμε το ε, δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δίνει το ε, παράδειγμα, να είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς. Αυτή η περίπτωση που βλέπουμε εδώ είναι χαρακτηριστική. Η Ήτρε δεν θα έπρεπε να είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και όχι μόνο για όλα αυτά ε, που ακούσαμε, αλλά και επειδή δεν είναι καθόλου αρμόδια για την σύσταση ενός τέτοιου ταμείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ομάδας EFTD, ο κύριο Καστάλιντο το Κύριος Καστάλιντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδέλφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, κύριο Μακάλιστερ για τις προσπάθειες που έκανε για τη σύνταξη αυτού του προσχεδίου. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως το EDIDP, το EDF δεν είναι μόνο ένα σημαντικό εργαλείο για την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει να προχωρήσουμε πραγματικά στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Μια συνεργασία ευρωπαϊκή πραγματική θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ε, τρία κράτη και τρεις επιχειρήσεις ε, ως μέλη. Κάτι που αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι βέβαιο έτσι όπως έχει διατυπωθεί το άρθρο 11.4. Μόλις πριν από λίγους μήνες αυτή η Επιτροπή και η Επιτροπή ΑΦΕΤ μετά από εντατικές συζητήσεις ε, επικύρωσε ότι ήταν το 3 3 σύστημα λογικό ε, για να υπερασπίσουμε τους ευρωπαϊκούς, ε, τις ευρωπαϊκούς στόχους. Το να είμαστε μυστικοπαθείς όχι μόνο θα μας απομακρύνει από μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά θα δημιουργήσει προβλήματα σε ένα ευαίσθητο θέμα που σήμερα χρειάζεται ενιαίο όραμα και ενιαίες προθέσεις. Διμερείς λογικές με αποκλεισμούς ε, και που δεν συμφωνούν θα μας απομακρύνουν από την νομική βάση του άρθρου 173 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα μπορέσουμε να αιτιολογήσουμε αυτή τη δαπάνη στον κόσμο. Και αυτό που αναφέρεται στο 12.1, ε, στο να υπάρχουν επιχορηγήσεις χωρίς έκκληση, δημιουργεί προβληματισμούς. Μια, ταυτόχρονη μια τέτοια συζήτηση έχει ήδη αναφερθεί, δημιουργώντας πολλές αμφιβολίες ε, ε, για την άμεση ανάθεση επιχορηγήσεων. Επίσης κάτι άλλο υπάρχει στο αρθρό 10. Εκεί αναφέρονται επιχειρήσεις ε, με έδρα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης αλλά με έλεγχο τρίτων χωρών. Είναι σημαντικές, ε, αναφέρονται, σημαντικές αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες υπό συνθήκης μπορούν να προσθέσουν αξία στην έρευνα και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων και τεχνολογιών στην Ένωση. Κάτι πιο πολιτικό τώρα οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα πρέπει να χρησιμεύουν στους τελικούς χρήστες. Με άλλα λόγια, δεν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας να μεταμορφωθεί σε ένα εργαλείο επιχορήγησης έμεσης της αμυντικής βιομηχανίας. Θέλουμε η στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη να βρει τη σωστή της θέση ώστε να αποφύγουμε επενδύσεις και αναπτύξεις προϊόντων που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι στρατιωτικοί μας. Η τεχνική λοιπόν οι τεχνικέ δυνατότητε των έργων θα πρέπει να συνάδουν με του τελικού χρήστε και τι ανάγκε τους. Σε αυτό επιμείναμε και χθε στην πολύ χρήσιμα συνάντηση με την ΕΝΤΑ. Το επαναλαμβάνω λοιπόν εδώ και το τονίζω, διότι ακούσαμε και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας τον ΙΔΕ ίδια οράματα και τις ίδιες προσπάθειες για συντονισμό βάσει των προτεραιοτήτων που έχουν εκφραστεί και όσον αφορά τα έργα τα οποία θα γίνουν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Αυτά ήταν κάποια κύρια θέματα που θα χαρακτηρίσουν τις τροπολογίες που θα υποβάλλω. Είμαι βέβαιος ε, ότι μαζί σας κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισηγητά, θα καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή έκβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη που υπήρξε εδώ μια παρεξήγηση, δεν ανημερώθηκα εν καιρά για τους σκιώδεις. Ε, ποιος θα την κυρία Βαλέρο, ο κύριος Κλωσμπούχνερ, λοιπόν, εκ μέρους των Πρασίνων, έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ και εσάς κύριε Μακάλιστερ για αυτήν την ε, πολύ καλή έκθεση. Όπως όλοι γνωρίζετε, καταψηφίσαμε αυτή την ρύθμιση για το ITP. Εμείς σε αυτήν την περίπτωση πιστεύουμε ότι 30 δισεκατομμύρια σε τομείς οι οποίοι δεν είναι αποτελεσματικοί δεν είναι κάτι που έχει νόημα. Για, για μας αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης Άμυνας δεν έχει και πολύ νόημα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετές ε, δομές. Το ταμείο αυτό θα προσθέσει μόνο στον καταγερματισμό των παρετέρω των 28 διαφορετικών ε, αμυντικών αγορών. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά για μας η πρόταση ενός τέτοιου ταμείου είναι ε, σαν να μας λείπει το θάρρος για να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά. Μια εσωτερική αγορά με κοινέ προδιαγραφές και πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι επειδή τα πράγματα έχουν όπως έχουν, χάνουμε 25 με 30 εκατομμύρια το χρόνο χρήματα των πολιτών. Πώς να εξηγήσουμε λοιπόν στον Ευρωπαίο φορολογούμενο ότι δεν θέλουμε να, να αλλάξει αυτή η δομή, αλλά αντίθετα θέλουμε να τους δίσουμε περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αυτήν την γνωμοδότηση θα επικεντρωθούμε στο να αποφύγουμε μια τέτοια σπατάλη για αυτά τα αυτόνομα όπλα, για το ουράνιο και για άλλη τεχνολογία. Και για μας θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά το έργο της Επιτροπής. Με την προπαρασκευαστική δράση για την αμυντική έρευνα βλέπουμε ότι είναι οι ίδιες επιχειρήσεις οι οποίες συμβουλεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή να μην υπάρχει πια αυτή η σύγκρουση συμφερόντων. Τέλος, κάνω έκκληση σε όλους σας να μην κάνουμε αυτό που έκαναν οι μεγάλες ομάδες στο EDIDP, να ελεγχθεί πρώτα καλά το πρόγραμμα εργασίας. Εδώ πρέπει να στηρίξουμε τις κατεξουσιοδότηση πράξεις για το πρόγραμμα εργασίας. Αλλιώς βοηθάτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει ένα από τα λίγα ε, στη δημοκρατία που δεν μπορούν να ελέγξουν αμυντικά προγράμματα. Δεν μπορεί να δίνουμε για 7 χρόνια επιταγή εν λευκό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος βουλευτής θα έκανε κάτι τέτοιο. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Κλέρ Μούντι, δεύτερη αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μακάλιστερ. Εξαιρετική γνωμοδότηση. Δεν μένουν και πολλά να προσθέσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός αναπόφευκτα. Ε, αλλά αναπόφευκτα πάντα μένει και κάτι βέβαια. Όσον αφορά τον προπολογισμό που αναφέρατε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. πρέπει πραγματικά να υπάρχουν τα απαραίτητα εχέγγυα να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα δαπανηθούν σωστά τα χρήματα αυτά. Αυτά που είπατε για την αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και αλλού και τα κενά θα πρέπει πραγματικά να συμπληρωθούν με αποτελέσματα συγκεκριμένα. Δεύτερον, έχουμε το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης. την ιδέα ότι δαπανώντας αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και τα πρότυπα εταιρική διακυβέρνηση. Ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει σε άλλα προγράμματα ε, όπως υπάρχει σε ένα αντίστοιχο σύστημα στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ε, όπου αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση στι ΗΠΑ για κάποιε εταιρείε που δεν πληρώνουν κάποιου κανόνε. Θα μπορούσαμε και εμεί να ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Μετά έχουμε την ε, αλυσίδα προμηθειών, ε, την αλυσίδα παραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείε αυτές, ξέρετε, είναι ειδικευμένες. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει ένα πιο λιγότερο περιοριστικό πρόγραμμα όσον αφορά την αλυσίδα παραγωγής ώστε να διασφαλίσουμε ότι πραγματοποιείται αποτελεσματική δαπάνη των κονδυλίων για να διασφαλιστούν τα αποτελέσματα που χρειάζονται και να λάβουν χρηματοδότηση και αυτές οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις επίσης. Η Κομισιόν αναφέρεται στην ε, συμβολή της ένταξης διαθέσεως του κλίματος μέσω της χρηματοδότησης. Αυτό αναφέρεται όμως και στη... δεν αναφέρεται ούτε στον κανονισμό, οπότε εμείς θα υποβάλουμε κάποιες ε, τροπολογίες για αυτή την ένταξη της διάσταση του κλίματος. Επίσης, όσον αφορά την ε, ισότητα των φύλων, έχω τελειώσει σχεδόν, σας το υπόσχομαι, προβλέπεται ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων στο Ταμείο και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν θα μιλήσω τώρα εκ μέρου όλων των συναδέλφων, αλλά ξέρω ότι γίνεται λίγο κουραστικό τελικά όταν κάθε κανεί μέσα σε μια τσέγγε ματιά, άντρε. Πολλέ γυναίκε ε, ε, κάνουν καριέρα σε αυτόν τον τομέα και μπορούν να συμβάλλουν ε, επικοδομητικά. Θα πρέπει λοιπόν να το αναφέρουμε. Και τέλο, ο κίνδυνος όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, όπως αναφέρεται στον κανονισμό Ε, τέτοια θέματα ε, εθνικής ασφάλειας να παρεμποδίζουν τον επαρκή έλεγχο από τον Όλαφ και αυτό είναι ένα εμπόδιο και θα πρέπει να το αναφέρουμε στον κανονισμό να υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής διεξαγωγής ερευνών και να είμαστε βέβαιοι ότι δεν πραγματοποιείται κατάχρηση ε, στον κανονισμό για να το πω έτσι του ρόλου της Όλαφ παρεμπόδιση του ρόλου του Όλαφ Κύριε Χίλντε Βάουτμαντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα συναδελφοί. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η στρατιωτική κινητικότητα έχει γίνει μεγάλη προτεραιότητα. Τη συζητήσαμε στο πρώτο σημείο, την ξανασυζητάμε τώρα και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το σωστό εξοπλισμό αλλά άλλο είναι να μπορούμε να αναπτύξουμε το δυναμικό μας στην κατάλληλη στιγμή και στον κατάλληλο χρόνο. Εξού και η σημασία της θεριωτικής κινητικότητας είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Οπότε, η διευκόλυνση για την Ευρώπη και τα 6,5 δισεκατομμύρια για την ε, στρατιωτική κινητικότητα είναι κάτι που χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή τον κύριο Καστάλντο το, για το έργο του. Συγγνώμη λέει κυρία Φωτήγκα, κυρία Βάτμαν, έχετε περάσει στο επόμενο σημείο, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ε, νόμιζα ότι συζητάγαμε τη δικιά σου έκθεση. Όχι, όχι, όχι, συζητάμε για το προηγούμενο. Για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Άμυνας του γνωμοδόση του κ. Μακάλιστερ. Μετά είναι το άλλο θέμα. Ο κύριο Αρνελίδη τώρα και εσεί αργότερα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μακάλιστερ, σας ευχαριστώ πολύ για τις προσθήκες και τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής, τις οποίες μας παρουσιάσατε σήμερα. Είμαι Γερμανός Ευρωβουλευτής του SPD και έχω τη στήριξη του Υπουργού Οικονομικών μας, ε, λέγοντας ότι μόλις ε, πρότεινε σε μια συνέντευξη του στη Γαλλία, στη Φιγκαρό, να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ε, οπλική βιομηχανία και οπλική αμυντική βιομηχανία. Ανακοινώθηκε ότι χρειάζεται ευρωπαϊκός πυλώνας ασφάλειας. Λοιπόν, στην Ένωση. Ωστόσο, η γερμανική αντιπροσωπεία έχει αρκετά προβλήματα με την πρόταση της Επιτροπής, ορισμένα από τα οποία ήδη αναφέραμε στις ε, διαπραγματεύσεις μας για τον κανονισμό DIDP. Καταρχάς, Θεωρούμε ότι ε, η απλή παροχή χρηματοδότηση για ε, θέματα άμυνας ε, δεν θα οδηγήσει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωση σε τομέα Άμυνα, ούτε και θα καταπολεμήσει τον κατακαιρματισμό στα κράτη-μέλη, τον οποίο έχετε ήδη αναφέρει και είναι πολύ εύστοχο επιχείρημα. Μετά, η αμυντική βιομηχανία διαφέρει από τις υπόλοιπες. Χρειάζεται ισχυρότερη πολιτική εποπτεία, κοινοβουλευτικό έλεγχο, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και αυτό σε όλα τα στάδια ε, της έρευνας, της ανάπτυξης, αλλά και ε, αξιολόγηση και παρακολούθηση. Και συμφωνώ με την ε, συνάδελφο που αναφέρθηκε σε αυτό. Μετά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εξαγωγές. Η Ευρωπαϊκή ε, οι διατάξεις που περιέχει το κείμενο δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, διότι θα έπρεπε να εξυπηρετούνται οι προτεραιότητες και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και, αυτή, και η πολιτική στρατηγική είναι προς το συμφέρον της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά δεν είναι το κέντρο αυτού. Θεωρούμε επομένως ότι ότι δεν είναι αρκετά ισορροπημένες ε, όλες οι διαστάσεις, ιδίως πολιτική και οικονομική. Μετά περνάω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο και να τονίσω ότι τα αυτόνομα οπλικά συστήματα δεν ε, είναι κάτι στο οποίο συμφωνεί το Κοινοβούλιο και πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είμαστε υπέρ των αυτόνομων οπλικών συστημάτων στην έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω πως ε, θα συζητήσουμε τα αυτόνομα οπλικά συστήματα σήμερα. Εδώ ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών και θα ήθελα να δώσω το λόγο ξανά στον David McAllister, τον εισηγητή της νομοδότησης. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, και τις συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θεωρώ ότι από κοινού μπορούμε να ε, πάμε την γνωμοδότηση σε πολύ καλό δρόμο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συμπεριλάβω όλες τις τροπολογίες σας ε, και να κάνω το καλύτερο μπορώ. Μία παρατήρηση επιτρέψτε μου. Δεν συμβαίνει συχνά να συμφωνούμε με την κυρία Λέζινγκ. Ε, το πολιτικό φάσμα στη Γερμανία είναι τεράστιο και οι διαφορές ανάμεσα στο δικό της κόμμα τη Λίνκε και το δικό μου το Τσεντεού είναι μεγάλο και αυτό θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η κυρία Λόζινγκ ε, έδειξε απίστευτη υπευθυνότητα και μπορώ να προσωπογράψω 100% αυτά που λέει. Ελπίζω να, ε, ελπίζω να μακάρι να είχαμε εμεί την αρμοδιότητα γι' αυτό. Όμω, η απόφαση που ελήφθη στην ε, διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών ήταν αυτή που είναι και το τι θα γίνει στη συνέχεια, αν θα προσφύγουμε εναντίον της απόφαση ή όχι, θα δείξει. Αυτή τη στιγμή όμως ε, και δεδομένου των γεγονότων νομίζω πως πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα μέσω της ε, γνωμοδότησης για αυτό το θέμα. Και θα υποβάλλω τις σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θεωρώ πως η αρμοδιότητα θα έπρεπε να μην είναι ε, στην Επιτροπή Τρέλα, στην ΑΦΕΤ και τη ΣΕΝΤΕ. Εδώ ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και όπως ε, είπε ο κύριος Μακάλιστερ προηγουμένως στις 5 Νοεμβρίου θα ψηφιστεί η έκθεση στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και στις 21 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Ίτρε. Η διαπραγματευτική εντολή για τον τριμερή διάλογο θα εγκριθεί το Δεκέμβριο, μάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. δημιουργία της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Η συγητής είναι ο κύριος Καστάλντο. Και μια και δεν έχουμε καθόλου χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Καστάλντο συνοπτικά να μας εξηγήσει την ε, διαδικασία ε, στην αρχή της παρουσίασης του, διότι πρέπει να βιαστούμε, δεν θέλουμε να χρονοτριβήσουμε τώρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ο μηχανισμός ε, συνδέοντας την Ευρώπη χρηματοδοτεί έργα για να καλύψουν τα κενά στα συστήματα της Ευρώπης μεταξύ ενέργειας, μεταφορών και ε, τα ευρυζωνικά συστήματα. Εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την άμυνα και την ασφάλεια που σημειώνει τεράστια επιτάχυνση και ε, αυτή τη στιγμή διαδίδεται ιδιαίτερα και στις συζητήσεις. Όσοι εισηγητής για τη συνεργατική κινητικότητα εδώ, ε, θέλω να αναφέρω τρεις γραμμές που έχουν χαρακτηρίσει τις τροπολογισμοί. Η πρώτη είναι το πλαίσιο στο οποίο επικεντρώνεται η στρατιωτική κινητικότητα από μόνη της δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς στενή συνεργασία με τη μη στρατιωτικό σκέλος. Ε, με άλλα λόγια, δεν θα ήταν οικονομικό να χρησιμοποιούμε, να κατασκευάζουμε υποδομές αποκλειστικά στρατιωτικές. Αντιθέτως, πρέπει να βρίσκουμε τους ε, μη στρατιωτικούς άξονες, ε, αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους κτλ. που μπορούν να χρησιμεύσουν και για στρατιωτικούς σκοπούς. Ε, οι υποδομές δηλαδή διπλής χρήσης με τις ανάλογες προσαρμογές ε, για τις στρατιωτικές ανάγκες αν χρειαστεί όλα αυτά λοιπόν να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα με το μη στρατιωτικό σκέλος με την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων με συμμετοχικές, αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες πιστεύω ότι η διπλή χρήση των υποδομών πρέπει να θεωρείται σημαντικό κριτήριο αναφέρομαι στα κριτήρια ε, ανάθεσης του αρθρού 13 τα στρατιωτικά πρότυπα μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω ασφάλεια στις εν λόγω υποδομές. Τέλος, η στρατιωτική κινητικότητα θα πρέπει να έχει προσοχή και σεβασμό προς την περιβαλλοντική διάσταση και στον τομέα της άμυνας. Όλα τα απαραίτητα πρότυπα για να διατηρηθούν οι στόχοι της Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Το δεύτερο θέμα είναι το γεωπολιτικό πλαίσιο που βρισκόμαστε σήμερα το τόξο κρίσης που χαρακτηρίζει την Ήπειρό μας ε, μας υποχρεώνει να επενδύσουμε με μακροχρόνιο όραμα αποφεύγοντας ε, συμφορήσεις στο μέλλον που μπορεί να επιβραδύνουν οποιαδήποτε αποτελεσματική κινητοποίηση η ε, επιχειρήσεις των στρατιωτικών μας δυνάμεων σε περίπτωση στρατιωτικής σύραξης αλλά και φυσικών καταστροφών. Τι σημαίνει αυτό ότι τα σημερινά μέσα δεν θα πρέπει να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον άλλες ε, προκλήσεις. Ε, τη στρατηγική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη γεωγραφική προσέγγιση και ισόρροπη. Θα πρέπει να επιτρέπεται εύκολη κίνηση ανθρώπων και υλικού ε, από το βορρά προς τον νότο όσο και στον άξονα Ανατολής Δύσης. Ε, στην ανάπτυξη περαιτέρω δυνατήτων δεν πρέπει να αξιολογούμε μόνο τις σημερινές προκλήσεις αλλά και τις ενδεχομένως μελλοντικέ σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, την ΠΕΣΚΟ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Το τρίτο είναι ότι η στρατιωτική κινητοποίηση δεν χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση κρίση. Αντιθέτω, χρειάζονται περαιτέρω περιθώρια παρέμβαση για εκρέμη ζητήματα, τελωνία, ε, διέλευση στρατιωτικών ε, αγαθών, εμπορευμάτων, ασφάλεια, μεταφορά γενικότερα αγαθών όπου συχνά οι κανόνες διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ώστε οι στρατιωτικέ επενδύσεις να αποδείξουν κάποια χρησιμότητα και σε περίπτωση ασκήσεων, αλλά και στην ε, ε, προώθηση υλικού σε περίπτωση ε, φυσικών καταστροφών ή για τη μετακίνηση των μέσων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνατότητες της στρατιωτικής κινητικότητας θα αποδώσουν αποτελέσματα σε μη στρατιωτικό και στρατιωτικό επίπεδο μόνο αν ε, είναι αλληλοσυμπληρωματικά ε, σε αυτές οι δύο διαστάσεις. Ευχαριστώ και τους Κιώδης και τους λοιπούς συναδέλφους για όλα τους τα σχόλια και με βέβαιο ότι θα καταφέρουμε να επιτελέσουμε μια επικοδομητική δουλειά όλοι μαζί. Ευχαριστώ. now I give the floor. Ευχαριστώ κύριε Καστάλντο. Δίνω το λόγο τώρα στον Σκιώδη του ΕΛΚ, τον Τίνο Ευχαριστώ πολύ κύριε Καστάλντο. Η γνωμοδότησή σας πιστεύω αποτελεί μια πολύ καλή προσέγγιση επικοδομητική, θετική. Όλοι συμφωνούμε με τα κυρία σημεία λέει ο κ. Κελάμ, και με βέβαιο ότι η διάσταση τη ασφάλεια για την ανάπτυξη μελλοντικών ευρωπαϊκών συνδέσεων ε, δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Πολλέ ε, αυτής αυτή τη ε, ε, διάσταση της ε, ασφάλειας και γενικότερα και της κυβερνοασφάλειας επίση πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η στρατιωτική κινητικότητα χρειάζεται συγκεκριμένα βήματα, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Ο κανονισμό των 6,5 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο τη ε, διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη είναι ένα πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι κοινέ ανάγκε. Θα πρέπει όμως να είμαστε ανοιχτοί και για περαιτέρω ε, ανάγκες. Αξιοποιώ λοιπόν την ευκαιρία αυτή είναι εδώ. Δράτω με τις ευκαιρίες για να απευθυνθώ και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη και να πω ας μην καθυστερήσουμε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που προβλέπονται διότι ο, καιρό, ο χρόνος πιέζει. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, όχι για τη δική σας γνωμοδότηση, αλλά γενικότερα Ελπίζω θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Το ζήτημα από τον κανονισμό τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, όλε οι δράσει αυτή τη διευκόλυνση έχει νόημα να είναι διπλή χρήση. Δεύτερον, τι θα κάνουμε με την προσέγγιση της Επιτροπής Τραν των εισηγητών εκεί που αναφέρονται σε δράσεις ε, που θα ήταν αποκλειστικά στρατιωτικές ε, ε, πάνω σε υπάρχουσες αστικές υποδομές. Αυτό θα απαιτεί κάποιο σχεδιασμό, κάποια έγκριση ή προγράμματα που έχουν ήδη προϋπολογισμό. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Και μετά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει οπωσδήποτε το ποσό του προπολογισμού να διατηρηθεί τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, ώστε να υπάρξει κάποια δυνατότητα βελτίωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων μα. Ευχαριστώ. κυρία από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καστάλτο για την πρότασή του όσον αφορά την τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής για τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Μπορούμε, πιστεύω εγώ, επίσης να βελτιώσουμε και κάποιες διαπιστώσεις γιατί οι ελπίδες της Επιτροπής Μεταφορών, τώρα είμαστε και είμαι στη ΣΕΝΤΕ βέβαια, αλλά συμμετέχω στην Επιτροπή Μεταφορών, πρέπει να δούμε μήπως και στα πλαίσια της διτής χρήσης μπορούμε να έχουμε κάτι θετικό στο πέρασμα των συνόρων, για παράδειγμα σιδηροδρομικά. Γι' αυτό θέλω να ασχοληθώ και με τη σημασία που έχουν οι κοινέ επιχειρήσεις που μπορούν να βοηθήσουν διασυνοριακά και να βοηθήσουν και την μη στρατιωτική πτυχή. Τώρα υπόθηκε και νωρίτερα όταν συζητήσαμε για τη στρατιωτική κινητικότητα ότι πρέπει να διευκρινίσουμε και θα το κάνουμε με την Γενική Διεύθυνση MOVE να δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση αυτή, γιατί ένα μέρος των 6,5 ε, δισεκατομμυρίων θα χρησιμεύσει στο blending, στο χρηματοδοτικό μείγμα που συνδέει το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην χρηματοδότηση. Εδώ Άρα είναι θέμα ρήτρα που υπάρχει στη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Τώρα για τις ε, συνέργειες. Όπως γνωρίζετε υπάρχει η πτυχή μεταφορές και εκεί μιλάμε για τη συνεργασία της ε, χρήσης μεταφορών, αλλά υπάρχει και η ψηφιακή πτυχή και η ενέργεια. Για το Κοινοβούλιο στο προηγούμενο, στην προηγούμενη διευκόλυνση συνδέοντας της Ευρώπης είχαμε μιλήσει για τη συνέργεια, γιατί η κινητικότητα και η στρατιωτική και η μη στρατιωτική χρειάζονται κάποια σύγκληση των τριών αυτών πτυχών. Μιλήσαμε για την κινητικότητα, συνδεδεμένη, η αυτόνομη. Χρειάζεται αυτή η σύγκληση. Τέλος, όσον αφορά την τροπολογία 11, μπορούμε και διμερώς βέβαια να το συζητήσουμε, αλλά επειδή προβλέπεται ήδη το θέμα της χρήσης, τα κονδύλια αυτά δηλαδή να χρησιμεύσουν αποκλειστικά για την διτή κινητικότητα, με τις δύο χρήσεις, δηλαδή στρατιωτική και μη στρατιωτική, ο περιορισμός που βάζετε εσείς μου φαίνεται εμένα σαν ένας διπλός περιορισμός και θα ήθελα να καταλάβω πού ακριβώς αναφέρεστε να δούμε ποιες θα έπρεπε να είναι οι προϋποθέσεις, οι εγγυήσει ώστε η χρήση να είναι πάντα δίτη χρήση και στρατιωτική και μη στρατιωτική. Θέλω να το καταλάβω καλύτερα. Γιατί έτσι φαίνεται σαν ένα παραπάνω περιορισμό σε κάτι που εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. για το μη στρατιωτικό τομέα δηλαδή, που μερικές φορές βρίσκεται πολύ πίσω. Πάντως είμαστε ικανοποιημένοι που υπάρχει δυνατότητα αυτής της διτής στρατιωτικής κινητικότητας γιατί μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο τους κύριους άξονες και τους δευτερεύοντες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε η πράσινη ο κύριος Κλάους Μπούχνερ εκ μέρους της κυρίας Βαλέρο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που θεωρώ μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είπαν σχεδόν όλοι, ότι δηλαδή τα προγράμματα όπως το συνδέοντας την Ευρώπη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ε, προγράμματα και έργα που αφορούν την Ένωση ευρωπαϊκά και όχι για εθνικά έργα ή για οτιδήποτε έχει σχέση με τον ΝΑΤΟ. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να διατίθεται σε ευρωπαϊκά project λοιπόν. Ε, ακούσαμε αυτές τις απόψεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να επεξεργαστούμε το κείμενο τόσο καλά έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε τέτοια χρήση θα υποβάλουμε ελάχιστε τροπολογίε, διότι νομίζω πω η έκθεση είναι μια πολύ καλή αφετηρία για ε, περαιτέρω δουλειά. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λυπάμαι πολύ που έχασα την, ε, ξέχασα την κυρία Βάουτμαν. Έχετε το λόγο. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Ναι, συνάδελφοι. όντω. Η στρατιωτική κινητικότητα, όπως είπα και στην αρχή, στο πρώτο θέμα που εξετάσαμε, είναι πάρα πολύ σημαντική και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καστάλτο και τον ευχαριστώ για το έργο του. Το είπαν όλοι οι συνάδελφοι ότι ε, συγχαρητήρια αξίζεται. Πρέπει να τονίσουμε ότι η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη αποτελεί ένα μέσο για βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, αλλά αποτελεί συγχρόνως και ένα μέσο για να ενισχύσει τη στατιωτική κινητικότητα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Καλά κάνουμε και κοιτάμε το θέμα συνολικά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Είναι πολύ καλό λοιπόν και πρέπει πράγματι να δούμε πώς συνδυάζονται όλα αυτά και με την ΠΕΣΚΟ με τη διαστρωμένη συνεργασία. Και εννοείται ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το τοπικό επίπεδο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό που κάπως μου λείπει και θα υποβάλω μία τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η στρατιωτική κινητικότητα είναι προς όφελος των πολιτών, προκειμένου οι πολίτες να κερδίσουν σε ασφάλεια. Και αυτό πρέπει να φανεί ότι θα προστατεύονται καλύτερα οι πολίτες. Είδαμε μετά τη Γένοβα. Οι επενδύσεις λοιπόν σε υποδομές είναι κάτι θετικό για τη στρατιωτική κινητικότητα, αλλά είναι καλό γιατί προστατεύονται έτσι καλύτεροι οι πολίτε και είναι και καλό και για την οικονομία. Συνεπώ, έτσι η Ευρώπη έρχεται πιο κοντά στον πολίτη και γίνεται περισσότερο ελκυστική. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καστάλτο, και σα είπα ότι θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καστάλτο, λόγο πάλι σε εσά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλου τους συναδέλφου ε, για τα πολύ ευγενικά τους λόγια για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Χαίρομαι που βλέπω ότι συμφωνείτε με την προσέγγιση. Είμαι πεπισμένος ότι θα καταφέρουμε να εργαστούμε γρήγορα, με συνένεση και με ακρίβεια. Τώρα, σύμφωνα με τη σειρά των παρεμβάσεων, εγώ σημείωσα φυσικά τα όσα είπατε. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Κέλαμ όταν λέει ότι το μήνυμα πρέπει να δώσουμε στην Κομισιόν να προσπαθήσει να τηρήσει τους χρόνους, δηλαδή να μην χάνουμε χρόνο άσκοπα σε αυτή τη σημαντική διαπραγματευτική φάση, να καταφέρουμε το συντομότερο δυνατόν να καταλήξουμε σε κάποια θετική έγκριση. Συμφωνώ επίσης ε, ότι είναι σημαντικό, όπως είπατε, το επίπεδο του προπολογισμού να διατηρηθεί, όπως είπατε, διότι μιλάμε για σημαντικό ποσό φυσικά, αλλά ξέρουμε και πόσο σημαντικές είναι και οι απαιτήσει. Ε, Αισθητέ, μάλιστα. Χαίρομαι που γενικότερα η προσέγγιση της διπλής χρήσης ε, ε, έχει υποστήριξη από όλους τους συναδέλφους. Ήθελα να διευκρινίσω κάτι γιατί μου το ρωτήσατε δύο φορές. Όσον αφορά την τροπολογία 11, αυτό που διευκρινίζεται όσον αφορά τα 6,5 δις, αυτά μπορούν να καλύψουν μόνο το κομμάτι του upgrade των, σε επίπεδο στρατιωτικών απαιτήσεων ε, σε μη στρατιωτική βάση. Αυτό εξηγεί αυτή τη στιγμή η πρόταση τη Κομισιόν που προσπαθώ να ξεκαθαρίσω, γιατί είναι σαφέ ότι αν αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια ήταν ολόκληρο το κόστο ε, ενό έργου διπλή χρήση, θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτύχουμε ευρεία κάλυψη. Αφού το ποσό είναι μεγάλο μεν, αλλά όχι απεριόριστο. Αυτή ήταν η πρόταση τη Κομισιόν. Αυτό προσπάθησα να ξεκαθαρίσω κατά κάποιο τρόπο αυτή την τυχή γιατί ήταν λίγο δυσνόητη η διατύπωση. Επίση, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που υπενθύμησε η συνάδελφο Ίνεσα Αγιαλά Σέντερ όσον αφορά τη δυνατότητα να σταματήσουμε αυτές τις επικρίσεις των διασυνεργατικών συνεργασιών ε, που μερικές φορές ε, αφορούν και επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να, να εξηγήσουμε ότι δεν υπάρχει λόγος για τόσο κριτική στάση και να ε, ξεκαθαρίσουμε τις αμφιβολίες. Η διευκόλυνση συνδέεται στην Ευρώπη έχει τρεις πυλώνες, ε, μιλάμε για, όπως είπατε. Καλό είναι να θυμίσουμε λοιπόν ε, και το θέμα όσον αφορά τις αστικές μεταφορές, όσο και τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές ε, με το TMS υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε που μπορούν να διασφαλίσουν και μεγαλύτερη συχνότητα ε, των δρομολογιών σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση πολλών γραμμών που, υπο, που πασχούν από υποεκμετάλλευση στον μη στρατιωτικό λοιπόν σκέλος να έχουμε όλα αυτά τα έργα αλλά να μην ξεχνάμε και τη στρατιωτική διάσταση η οποία μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για πιο γρήγορη εφαρμογή. Ε, να βελτιωθούν κάποιο ποσοστά από αυτή τη στιγμή είναι χαμηλά. Είδα ότι γενικότερα συμφωνούμε ευρέως ε, ε, για την ανάθεση των κονδυλίων και των γενικών και των ειδικών. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφός κ. Μπουκνέρ. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια. Σίγουρα θα εστιαστούμε με το Συνδέοντα στην Ευρώπη στι ευρωπαϊκέ αξίε και στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ναι, φυσικά πρέπει να υπάρχει κάποιο βαθμό συντονισμού μεταξύ των διαφορών πτυχών και των κρατών και των προγραμμάτων, αλλά εμεί είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτά τα χρήματα θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ε, που θα χρησιμοποιηθούν για προσθεμένη αξία ευρωπαϊκή, αποφεύγοντας επικαλύψεις ε, ή να γίνουν παρεμβάσεις που έχουν ήδη προβλεφθεί αλλού, πάντα σε πλαίσιο συνέργειας φυσικά και με πάντα γνώμονα την προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Βάουτμαντς. Συμφωνώ, απαιτείται να συντονιστούμε φυσικά και με την ΠΕΣΚ. Το συζητήσαμε και χθε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα ε, στο γεύμα εργασία που είχαμε. Ε, προχωράει η διαδικασία εκεί. Ε, για το ετήσιο πρόγραμμα με τους στόχους και τις ανάγκες ε, που πρέπει να επιδιώξουμε και προφανώς ε, είμαι πολύ ικανοποιημένος που αναφερθήκατε στη συμμετοχή των τοπικών οργανισμών, των τοπικών κοινοτήτων αρχών του υποεθνικού επίπεδου ώστε τα προγράμματα αυτά να βρίσκουν όλους σύμφωνους ε, να έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση με άπαντες και να θεωρούνται ε, από τις τοπικές κοινότητες ως κάτι θετικό, ως ε, Και γι' αυτό εστιάζουμε και στη βιωσιμότητα. Είναι σαφές ότι το να γίνεται μια αναβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων σημαίνει ότι αναβαθμίζονται γενικότερα οι συνθήκες ασφάλειας. Και φαντάζεστε ότι εγώ ως Ιταλός και μην ξεχνώντα την τεράστια τραγωδία που έλαβε φέτο το καλοκαίρι χώρα στην ε, Γιάνοβα, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για μένα αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Είμαι πεπισμένο ότι αν χρησιμοποιήσουμε σοφά και συνεργατικά τα χρήματα αυτά έτσι όπως το προτείνουμε θα μπορέσουμε να επιτύχουμε καταπληκτικού στόχου με εξορθολογιστική χρήση των δαπανών και έχοντα υπόψη μα ότι θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να χρησιμοποιηθούν από κοινού για τη δική μας ασφάλεια και άμυνα αλλά και προς το συμφέρον των πολιτών μας που τελικά θα πρέπει να τα δουν όλα αυτά ως μια ευκαιρία και όχι ως μια απομακρυσμένη ε, θεματολογία σε σχέση με την καθημερινότητά τους. Χαίρομαι που θα συνεργαστούμε. Πρόεδρε, συγγνώμη πρέπει να σας διακόψω γιατί είμαστε, έχουμε καθυστερήσει το πρόγραμμα. Συνάδελφοι, Λυπάμαι πολύ, αλλά πρέπει να ολοκληρώσω τη συζήτηση για αυτό το σημείο. Ε, γνωρίζω πω ε, επιθυμούν να λάβουν και άλλοι συνάδελφοι το λόγο, όμω δεν μα φτάνει ο χρόνο και έχουμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό θέμα με ανταλλαγή απόψεων να εξετάσουμε. Και έχουμε και εξωτερικού προσκεκλημένου Είμαστε ευγνώμονες ε, στον κύριο Καστάλντο γιατί ανέλαβε αυτήν την ε, επικίνδυνη αποστολή. Δεν έφτανε ο χρόνος, οι ε, αρμόδιες επιτροπές, η Ήτρε δηλαδή και η Τραν δεν μας άφησαν καθόλου χρόνο, οπότε ήταν πολύ θαραλέος ο κύριος Καστάλντο που το ανέλαβε. Τροπολογίες στις 11 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι. Δεν θα ε, επαναξετάσουμε το θέμα και επίσης ε, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ θα εγκριθεί το σχέδιο έκθεση 27 Σεπτεμβρίου. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν κύριε Καστάλιντο για την παρουσίαση. Προσβλέπουμε στο τελικό κείμενο και σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον των αυτόνομων όπλων. Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τους ε, εκλεκτούς προσκεκλημένους μας, τον κύριο Μάικλ Κάλεντερ, επικεφαλής στον τομέα αεροδιαστημικών ικανοτήτων του ΝΑΤΟ και την κυρία Ουλρίκη Έστερ Φράνκε, είναι συνεργάτητα σε θέματα πολιτικής ε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Δεν θέλω να σπαταλήσω λοιπόν άλλο χρόνο γιατί το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και ενδιαφέρον και όλοι θέλουμε να το συζητήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας χωρίς καμία καθυστέρηση. Κύριε Φράγκη, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσετε. Έχετε το λόγο, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα για να μιλήσω για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, το μέλλον δηλαδή των αυτόνομων όπλων. Στόχος μου σήμερα είναι να σας δώσω μια γενικότερη εικόνα της τεχνολογίας, των ε, ζητημάτων και της ε, κατάστασης της ε, συζήτησης για τα ρομπότ έτσι όπως λένε τα θανατηφόρα αυτόνομα όπλα. Είναι πολύ καλή χρονική στιγμή για αυτή τη συζήτηση, διότι την περασμένη εβδομάδα στην Γενέβη εκπρόσωποι πάνω από 70 χωρών, με συγχωρείτε, διακόπτη πρόεδρος, Συνάδελφοι, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε από την αίθουσα, παρακαλώ να το κάνετε με ησυχία. Να είστε ήσυχοι, θέλουμε ησυχία. Μας ενοχλείτε. Σας ευχαριστώ. Όπως έλεγα λοιπόν, είναι κέριο το... κέρια χρονική στιγμή, διότι όπως γνωρίζετε στη Γενέβα την περισμένη εβδομάδα συναντήθηκαν εκπρόσωποι από πάνω από 70 χώρες στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, φυσικά και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συζητήσουν το θέμα αυτό. Και με μεγάλη μου χαρά θα σας ενημερώσω για την πορεία των συζητήσεων στις ερωταπαντήσεις αργότερα. Να ξεκινήσω όμως ε, με το τι είναι τα θανατηφόρα αυτόνομα όπλα, γιατί αναπτύσσονται και γιατί ορισμένοι ζητούν την ε, απαγόρευσή τους. Σύντομα λοιπόν, lethal autonomous weapons, LOS, Αυτά είναι όπλα τα οποία μπορούν να εντοπίσουν και να καταστρέψουν στόχους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. αυτό είναι έτσι ένα σύντομος και σαφής ορισμός, όμως όπως ε, συνηθίζεται στις λεπτομέρειες είναι το ζουμί. Ε, να σας ε, δώσω δηλαδή μια εικόνα. Η αυτονομία δεν είναι κάτι σταθερό και σίγουρο, δεν είναι ένα όπλο αυτόνομο ή όχι, είναι ένα φάσμα και καθώς προχωράει η τεχνολογία, ιδιαίτερα καθώς προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη, ε, μετακινούμαστε μέσα στο φάσμα προς μεγαλύτερη αυτονομία. Στο ένα άκρο του φάσματος ε, ε, έχουμε την περίπτωση του ξελοθρευτή από την ταινία. Ένα FES θανατηφόρο ρομπότολοφόνος όπως ξέρουμε και από τις ταινίες. Από την άλλη μεριά του φάσματος όμως υπάρχουν συστήματα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται σήμερα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο γερμανικός στρατός χρησιμοποιεί τα συστήματα αεράμινας Μάντης και πάτριο. Αυτά τα συστήματα εντοπίζουν, παρακολουθούν και καταρρύπτουν ε, εισερχόμενους ε, πυράβλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο κέντρο ελέγχου και πατάει το κουμπί για κάθε ε, ενέργεια, κάθε εντοπισμό. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άλλο το αυτόματο και άλλο το αυτόνομο. Τα αυτόματα συστήματα ε, δεν λαμβάνουν τα ίδια αποφάσει, είναι προγραμματισμένα για να κάνουν συγκεκριμένε ενέργειε. Άλλο σύστημα, ε, το σύστημα Harpy στο Ισραήλ ή Harop, είναι ένα σύστημα όπως λέμε fire and forget, το οποίο δημιουργεί, χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό και εντοπίζει ε, εκπομπές ε, ραντάρ καταστρέφει αυτά τα ραντάρ ε, προσκρούοντας ε, στη, στον πομπό. Και κατά μία έννοια το σύστημα αυτό αποφασίζει να επιτεθεί όχι σε ένα ραντάρ. Όπως βλέπετε λοιπόν, ε, το να καθορίσουμε τι είναι αυτόνομο και τι όχι είναι κάπως δύσκολο και αυτή τη στιγμή υπάρχουν συστήματα τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό του αυτόνομου σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι τα αυτόνομα όπλα είναι εκείνα που λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε βάθος χρόνου και με δυναμικό ε, μη ε, ε δομένο ανοιχτό περιβάλλον. Μία κινητή πλατφόρμα χρησιμοποιεί ε, και ε, αλγόριθμους που του επιτρέπουν στο σύστημα αυτό να λάβει αποφάσεις και να τις εκτελέσει. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Υπάρχει μια σημαντική σύνδεση ανάμεσα στην αυτονομία και την τεχνητή νοημοσύνη, παρότι δεν είναι το ίδιο. Η νοημοσύνη, ε, μιλώντας ε, για έναν υπολογιστή, τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν, είναι η δυνατότητα ενός συστήματος να καθορίσει την καλύτερη ε, δράση έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του. Η αυτονομία όμως είναι η ελευθερία που έχει ένα σύστημα να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Για παράδειγμα, η λιγότερη εποπτεία σημαίνει περισσότερη αυτονομία. Και για να γίνει ένα σύστημα πιο αυτόνομο θέλεις και να είναι πιο ευφυές. Είναι όμως απόλυτα δυνατό να υπάρχει ένα ιδιαίτερα ευφύ σύστημα με ελάχιστη αυτονομία. Τι κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή και τι υπάρχει ήδη. Η Human Rights Watch ε, αναφέρει ότι η Κίνα, το Ισραήλ, η Ρωσία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείε αναπτύσσουν τέτοια αυτόνομα ε, θανατηφόροπλικά συστήματα. Λόγος από εδώ και στο εξή. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν δηλώσεις και να, και να πούμε με σαφήνεια τι κάνει, ποιος κάνει τι. Ορισμένα κράτη ενεργούν υπό απόλυτη μυστικότητα, άλλα από την άλλη... Ε, το δηλώνουν και όλα και είναι περήφανα γι' αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να δούμε απ' έξω τι ε, δυνατότητες έχει ένα σύστημα και αν ένα σύστημα είναι αυτόνομο ή όχι, διότι η αυτονομία έχει να κάνει με το λογισμικό και όχι το υλικό. Αυτό φυσικά δημιουργεί ε, προβλήματα στους μηχανισμούς ε, ελέγχου των όπλων και ένας άλλος λόγος ε, για τον οποίο είναι δύσκολο να δούμε ποιος κάνει τι, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι οι περισσότερες καινοτομίες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης δεν γίνονται από κρατικά ή στρατιωτικά όργανα, αλλά από πανεπιστήμια, εταιρείες, από ε, πολιτικούς οργανισμούς δηλαδή και ερευνητικά ιδρύματα. Όμως, ε, τι γίνεται στην Ευρώπη, μιας και είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα αναφερθώ στο βρετανικό ταράνις και στο γαλλικό ε, πανευρωπαϊκό neuron ε, σύστημα, τα συστήματα drone. Και τα δύο είναι μία επανδρομένα μαχητικά αεροσκάφη, δηλαδή οπλισμένα drones, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο επίδειξης. Είναι μία απόδειξη ψηλά ε, αυτόνομων συστημάτων, τα οποία ξεκίνησαν το 2005 να αναπτύσσονται, έχουν συμπληρώσει αρκετές δοκιμαστικές πτήσεις και στόχο έχουν ε, αναγνωριστικές πτήσεις, αυτόνομη πτήση και αναγνώριση στόχων, ε, όλα αυτά λειτουργώντας υπό αυτονομία. Αυτά τα συστήματα θα είναι ιδιαίτερα αυτόνομα, θα έχουν τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να απογειώνονται και να προσγειώνονται αυτόνομα, να διενεργούν αναγνωριστικές πτήσεις, έρευνες, να, να εντοπίζουν στόχους και το γαλλικό ευρωπαϊκό σύστημα Neuron έχει χαρακτηριστεί το, το σύστημα με την περισσότερη αυτονομία ε, στον κόσμο από την ε, βάση δεδομένων Global Security Initiative. Είναι μια βάση δεδομένων στην Αριζόνα που εξετάζει αυτή τη στιγμή 283 απλικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή ούτε το Ταράνις ούτε το Neuron δεν ε, προγραμματίζεται να εντοπίζουν στόχους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, όμως αυτό δεν, δεν απέχουν πολύ από το να το ε, κάνουν. Το θέμα είναι αν υπάρχει επαρκής ανθρώπινος έλεγχος. Και να σας ε, παρουσιάσω για ποιο λόγο αναπτύσσονται και κατασκευάζονται αυτά τα οπλικά συστήματα Λόγος Από στρατιωτική ε, οπτική, αυτά τα αυτόνομα θανατηφόρα όπλα προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα. υπόσχονται νέες στρατιωτικές ικανότητες και, μειωμέ, και μειωμένες ανάγκες ανθρώπινο δυναμικό ταχύτητα, είναι πολύ πιο γρήγορα τα οπλικά αυτά συστήματα από τους ανθρώπους και λέγεται ότι ο πόλεμος ε, μάλιστα στο μέλλον θα είναι υπερβολικά γρήγορος ε, από ε, την δυνατότητα των ανθρώπων να λάβουν αποφάσεις. Ιδιαίτερα αν η μία πλευρά χρησιμοποιεί αυτόνομα συστήματα. Μετά, stealth. Είναι πολύ σημαντικό να μην εντοπίζεται ένα σύστημα ε, ένα drone για παράδειγμα. Διαφέρει πάρα πολύ από ένα επανδρομένο όχημα, διότι ο πιλότος πρέπει να έχει κάποια επαφή με ένα κέντρο ελέγχου. Αυτές οι επαφές είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν και να αποκαλύψουν ε, μάλιστα πολλές φορές την τοποθεσία ε, από την οποία εκπέμπουν. Το αυτόνομο σύστημα όμως λειτουργεί σε δυνατότητα απόκρυψης και δεν μπορεί να εντοπιστεί. Τα συστήματα αυτά επίσης είναι πιο αποτελεσματικά διότι έχουν περισσότερη ακρίβεια στο Τα συστήματα αυτά μπορούν να διακρίνουν με μεγαλύτερη ευκολία ανάμεσα σε ε, στόχους αμάχων και στρατιωτικούς στόχους ε, και στόχος επίσης είναι να δημιουργήσουν νέες στρατιωτικές δυνατότητες. Τα σμήνι είναι η λέξη κλειδί. Swarm. Αυτά θα αποτελούνται από αρκετές ε, δεκάδες ή και εκατοντάδες τέτοια drones, πολλές φορές και χίλια τέτοια αυτόνομα οχήματα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτή η αυτονομία έτσι ώστε το Σμήνος να αναλάβει μία εντολή και να μπορεί να συντονιστεί το ίδιο για το πώς θα την εκτελέσει. Αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές έρευνες για τα Σμήνη μη επανδρομένων ε, οχημάτων στις Ηνωμένε Πολιτείε ιδιαίτερα. Και Τέλο, είναι ελκυστικά τα αυτόνομα συστήματα διότι μειώνουν τι ανάγκε ανθρώπινο προσωπικό. Οι στρατιώτε δεν θα χρειάζεται να μπουν σε πόλεμη και επικίνδυνη ζώνη, θα στείλουν τα ρομπότ δηλαδή. Τα αυτόνομα όπλα μειώνουν το σωματικό ε, και πνευματικό φόρτο για τους, ε, που χρειάζεται από τους στρατιώτες και όταν υπάρχουν και λιγότεροι στρατιώτες θα ε, μειώνεται και η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Όμως, να κλείσω την παρουσίασή μου λέγοντας ότι φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα που συνεπάγεται η χρήση αυτών των ε, συστημάτων και γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνει ε, συζήτηση. Γι' αυτό και ζητούν ε, πολλές ομάδες την απαγόρευση αυτών των αυτόνομων οπλικών συστημάτων. Θα περιοριστώ στις ερωτήσεις τεχνικού, πολιτικού και ε, ηθικού χαρακτήρα, διοντολογία και θα ε, περιοριστώ μόνο στα νομικά από αυτά. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτό που λέμε μαύρα κουτιά. Τι σημαίνει αυτό. Τα συστήματα που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη δεν ε, είναι προγραμματισμένα, αλλά έχουν μάθει. Έχουν μάθει με διάφορους τρόπους και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είναι πλέον σε θέση να κατανοήσουν απόλυτα το σκεπτικό και τη λογική του μηχανήματος. Αυτό τι σημαίνει όμως. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε τα λάθη που θα κάνει μια, ένα τέτοιο μηχάνημα. Και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο κάνουν λάθη, αλλά τα λάθη αυτά είναι και περίεργα. Κάνουν λάθη τα οποία δεν θα έκανε ποτέ άνθρωπος. Για παράδειγμα, ένα μηχάνημα μπορεί να εντοπίσει ένα τεθωρακισμένο 10.000 φορές σωστά. Όμως, την επόμενη φορά θα δει κάτι που θα θεωρήσει τεθωρακισμένο και θα είναι πεπισμένο το σύστημα ότι αυτό είναι τεθωρακισμένο, αλλά ε, μπορεί να είναι, το σύστημα θα νομίζει πως είναι κάτι άλλο, πως είναι μια γάτα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν για τους ανθρώπους να καταλάβουν για ποιο λόγο αυτά τα αυτόνομα συστήματα μπορεί να κάνουν λάθος. Και τώρα που μιλάμε για λάθη, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και συχνά είναι προκατηλημένη. Ίσως σας φανεί περίεργο αυτό, διότι έχουμε συνηθίσει τους οι υπολογιστές, 100% πιθανότητες ε, δεν, κάνουν λάθος. Όμως, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ε, ξέρουν τόσα όσα τους έχουμε προγραμματίσει να μάθουν. Και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά γενικά την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο τα αυτόνομα οπλικά συστήματα. Οι αλγόριθμοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών των Ηνωμένων Πολιτειών δοκίμασε αυτά τα συστήματα αναγνώρισης εικόνας που, χρησιμοποιούν τα, που χρησιμοποιεί η αστυνομία, τον είπα. Και σύγκρινε φωτογραφίες από βουλευτές του Αμερικανικού Κογκρέσου ε, με μία βάση δεδομένων ε, φωτογραφιών από εγκληματίες. Και το σύστημα λοιπόν τι έκανε, ε, ταύτισε 28 βουλευτές Αμερικανούς με εγκληματίες που έχουν συλληφθεί. Και αυτές οι, αυτά τα λάθος μάτς λοιπόν ε, μάλιστα ήταν ε, ιδιαίτερα για ε, έγχρωμους ε, ανθρώπους, αφορούσαν έγχρωμους ανθρώπους. Τελευταίο τεχνικό πρόβλημα είναι βάλατα τα συστήματα αυτά διότι μπορούμε να τα εξαπατήσουμε. Όπως και ένα σύστημα μπορεί να περάσει ένα τεθωρακισμένο για μια χάτα, έτσι μπορούν να γίνουν και άλλα λάθη. hacker μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ε, αδυναμία για να σαμποτάρουν τα συστήματα. Και όπως είπα, όποιος χρησιμοποιεί ένα τέτοιο σύστημα δεν θα είναι σε δυνατότητα να το κατανοήσει πλήρως και αυτό συνεπάγεται και ότι δεν θα είναι σε δυνατότητα να εντοπίσει ένα χακάρισμα που θα γίνει. Επίσης, πολιτικά υπάρχουν και πάρα πολλές ανησυχίες σχετικά με αυτά τα αυτόνομα συστήματα. Ε, η κυριότερη είναι ο φόβος ε, του ότι η ύπαρξη και μόνο αυτών των ε, δολοφόνων, των ρομπότ δολοφόνων θα πυροδοτήσει μία κούρσα για τα όπλα. Υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος κλιμάκωσης της κατάστασης, διότι τα συστήματα αυτά έχουν αυτό το πλεονέκτημα ταχύτητας που αναφέρα νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν είναι και λογικό ακόλουθο αν μια χώρα ξεκινήσει με την ε, χρήση αυτών των συστημάτων να ακολουθήσουν και άλλες. Τέλος, συστήματα δεοντολογίας. Και κλείνω με αυτό, διότι θεωρώ πως αυτά τα ζητήματα, τα ηθικά ζητήματα, είναι τα πιο σημαντικά ε, στο πλαίσιο όλης της συζήτησης και γι' αυτό θεωρώ πως το κοινό πρέπει να είναι ενημερωμένο. Θα έλεγε κανείς ότι τα ρομπότ δεν μπορούν να ε, εκτιμήσουν την αξία της ανθρώπινης ζωής και την απώλεια αυτής. Ε, θα παίρνουν αποφάσεις ζωή και θανάτου βασισμένα σε αλγόριθμους και οι ανθρώπινες ζωές ε, δεν θα είναι τίποτα άλλο από στόχοι. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτά παραβιάζουν την, τις αρχές της ίδιας ανθρωπότητας. Δύσκολο θα είναι βέβαια να πάρουμε μια απόφαση τώρα, όμως τα θα πρέπει εμείς να αναρωτηθούμε ως άνθρωποι, ως το σύνολο της ανθρωπότητας, ε, αν θα έπρεπε να αφήσουμε τους υπολογιστές να λαμβάνουν αποφάσεις ε, για τη ζωή μας, ερήμην μας. Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσει η κοινωνία στο σύνολό της και γι' αυτό περισσότερο μάλλον γι' αυτό παρά για οτιδήποτε άλλο είναι πολύ σημαντικό να ε, συζητηθεί το θέμα. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο έγινε συζήτηση στη Γενέβη την περισμένη εβδομάδα και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ ε, με το ότι εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή σας ε, ε, κάνετε αυτή τη συζήτηση για να ακούσετε τις απόψεις και κλείνοντας θα σας ευχαριστήσω ακριβώ γι' αυτό. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον Μάικλ Κάλεντερ. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Μάικλ Κάλεντερ και είμαι επικεφαλής ε, της αεροδιαστημικής ικανότητας ε, στα πλαίσια των αμυντικών επενδύσεων του ΝΑΤΟ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Τα σχόλιά μου πιστεύω ότι έρχονται πολύ καλά μετά από αυτά που ακούσαμε από την Δ. Φρέγκε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να έχουμε ίσως περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις αργότερα, ώστε να διαφωτιστείτε καλύτερα για αυτά που θέλετε να μάθετε. Ε, προειδοποιώ τους διερμηνείς, λέω μιλητής, ότι μιλάω γρήγορα, οπότε αν το παρακάνω, κάντε μου νόημα. Λοιπόν, ως επικεφαλής της αεροδεστημικής ικανότητας ε, του ΝΑΤΟ, θέλουμε να ενσωματώσουμε όσο γίνεται καλύτερα τα χερσαία συστήματα, δηλαδή τα συστήματα παρακολούθησης εδάφους καλύτερα του ΝΑΤΟ. Βέβαια, όταν μιλάμε για αυτονομία, αυτό είναι μια ψευδέστηση, γιατί πρόκειται για ένα σκάφος που έχει μια αυτοματοποιημένη ικανότητα, αλλά υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στον πιλότο και το σκάφος. τι θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο αυτόνομο σύστημα. Να ξέρετε ότι ένα οπλικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζει μια προσπάθεια. Ένα οπλικό σύστημα δηλαδή μπορεί να είναι από ελικόπτερο μέχρι ένα σκάφος μεταφοράς, οτιδήποτε. Στην περίπτωση λοιπόν των περίφημων συστημάτων παρακολούθησης εδάφους, πρόκειται για μια πλατφόρμα αναγνώρισης που δεν φέρει όπλα, δεν είναι εξοπλισμένη με οπλικά συστήματα. Μιλάμε όμως για ένα αυτόνομο οπλικό σύστημα παρόλα αυτά. Γενικά μιλώντας, όταν μιλάμε για αυτονομία και για ένα αυτόνομο οπλικό σύστημα, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορεί να επιλέξει τη διαδρομή του βάσει ενός προγράμματος που έχει ενσωματωθεί σε αυτό προηγουμένως χωρίς την ανθρώπινη ανάμιξη. Αλλά πρόκειται για προγραμματισμένα σχέδια πτήσης ουσιαστικά και τίποτα άλλο, δεν πρόκειται για αυτονομία. Οπότε θα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή μια επιλογή. Αυτή η επιλογή βασίζεται σε μία παλέτα ε, προγραμματισμού που έχει ενσωματωθεί στο μηχάνημα. Είναι λιγάκι σαν τα νέα συστήματα cruise control που έχουμε στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα, τα οποία προσαρμόζονται. Μπορεί να μην είναι η παρομοίωση τέλεια, αλλά παρόλα αυτά ε, λέμε ότι πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη ταχύτητα το σύστημα cruise και συγχρόνως όμως να κρατάει μια απόσταση από το αυτοκίνητο που προηγείται. Όλα αυτά τα έχει συνσωματώσει προηγουμένω στο σύστημα. Κάπως έτσι πρέπει να σκεφτούμε και την αυτονομία αυτή που βρίσκεται στα συστήματα παρακολούθησης εδάφους της συμμαχίας. Έχει βέβαια ένα περίπλοκο προγραμματισμό. Λειτουργεί όμως ε, από κάποιον πιστοποιημένο πιλότο διότι οι κανόνες, οι ρυθμίσεις που έχουμε καθαρίσει για τέτοιες ε, πτήσεις είναι ότι πρέπει να μπορεί να βλέπει και να αποφεύγει το σκάφος κάτι ενδεχομένω. Πρέπει να υπάρχει μια τακτική αποφυγής και για αυτήν φροντίζει ο πιλότος, ο οποίος βλέπει και μπορεί να κατευθύνει από μακριά το αεροσκάφος ώστε να διατηρήσει την απόστασή του όπως πρέπει από κάποιο εμπόδιο ας πούμε. Οπότε μπορεί να κάνει πολλά το αεροσκάφος και μπορεί να πάρει αποφάσεις, όμως ο πιλότος βρίσκεται από την άλλη μεριά βρίσκεται στο έδαφος και έχει επικοινωνία τελικά με το μηχάνημα αυτό. Δεν καθορίζει δηλαδή το σύστημα παρακολούθησης εδάφους από μόνο του το ποια θα είναι η αποστολή του, αλλά ακολουθεί μια πτήση βάση ενός προγραμματισμού. Τώρα για να είμαστε πιο ακριβείς, πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο έχει κάποιες λειτουργίες οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα με τη βοήθεια όμως ενός πιστοποιημένου πιλότου. Δεν παίρνει αποφάσεις από μόνο του. Δεν πρόκειται για ένα σύστημα εκτοξεύω και ξεχνάω. Απαιτεί την ανάμειξη του ανθρώπου σε διάφορα σημεία όπου πρέπει να πάρει μια απόφαση. Πότε πρέπει να προσγειωθεί. Για παράδειγμα, αποφασίζει ο πιλότος γι' αυτό. Για να είναι πραγματικά αυτόνομα ένα τέτοιο σύστημα και το ανέφερε και η δόκτωρ Φράγκε και είναι πολύ σωστό και σημαντικό αυτό στη συζήτηση, σημαίνει ότι πρέπει να έχει την ικανότητα να δράσει σύμφωνα με τους δικούς του στόχους, τις δικές του αντιλήψεις, τη δικιά του κατάσταση χωρίς εξωτερική παρέμβαση και να βασίζεται μόνο στις δικές του ανιχνευτικές ικανότητες. Και αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που μπορεί να κάνει το σύστημα παρακολούθησης εδάφους της συμμαχίας. Και γιατί γιατί η τωρινή πολιτική του ΝΑΤΟ για τα μη επανδρομένα αεροπορικά συστήματα είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ το ΝΑΤΟ. Σημαίνει ότι δεν είναι επανδρομένα και ότι μπορούν να λειτουργήσουν με κατεύθυνση από μακριά. Το ΝΑΤΟ δεν έχει μία πολιτική αυτόνομων αεροσκαφών και όπως εξήγησε η Δ. Φράνκε μπορεί να το θελήσουμε κάποια στιγμή και η τεχνολογία σίγουρα προδεύει και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς. Αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να συμφωνήσουν και να ζητήσουν από τον ΝΑΤΟ να αναπτύξει μια τέτοια πολιτική. Αυτό ισχύει λοιπόν και για αυτόνομα ε, συστήματα οπλικά. Πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες για κάτι τέτοιο. Πρέπει να πούνε στο ΝΑΤΟ να αναπτύξει μια τέτοια πολιτική αυτόνομων οπλικών συστημάτων. Βέβαια το ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την τεχνολογία αυτή αυτόνομων οπλικών συστημάτων. Η κοινοτομία όμως ε, βασίζεται περισσότερο στον εμπορικό τομέα και όχι στον στρατιωτικό όπως είπε και ο Δ. Οι συνολικές ε, επενδύσεις που γίνονται από τις κυβερνήσεις κυρίως είναι βέβαια σημαντικές. Η αυτονομία λοιπόν βασίζεται στις έρευνες που γίνονται στον εμπορικό τομέα. Οι συνολικέ επενδύσει το 2014 ήταν τρισεκατομμύρια εκατομμύρια δολάρια επενδύσει στην πληροφορική. Οι συνολικέ στρατιωτικέ ε, ε, δαπάνε για τη ρομποτική είχε προβλεφθεί για φέτο να είναι 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να συγκρίνουμε, οι συνολικές δαπάνες βιομηχανικές και εμπορικές στη ρομποτική εκτιμήθηκαν στα 43 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Βλέπετε λοιπόν τη σύγκριση των στρατιωτικών δαπανών με τις βιομηχανικές και τις εμπορικές. Θέλω να πω ότι την καινοτομία την κάνει ο βιομηχανικός και εμπορικός τομέας και όχι ο στρατιωτικός. Το ΝΑΤΟ βέβαια ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά και θέλει να ενημερώνεται. Έχουμε 5.000 επιστήμονες που ασχολούνται με 250 επιστημονικές δραστηριότητες στο ΝΑΤΟ, έτσι, για να ενημερώνονται για τις εξελίξεις. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι 250 αυτές επιστημονικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν ε, απευθείας με την ε, ε, τεχνητή νοημοσύνη. Όμως ή την αυτονομία των συστημάτων, όμως μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τι υπάρχει, τι δυνατότητες υπάρχουν και τι χρειάζεται για να γίνουν πραγματικότητα αυτές. Θέλουμε να ξέρουμε τι κάνουν οι χώρες μέλη και τι κάνουν και οι εταίροι του ΝΑΤΟ. Τώρα το θέμα της ε, αυτονομίας και των αυτόνομων συστημάτων δεν είναι μόνο επιστημονικό ζήτημα, έτσι. Γιατί τι κάνει τελικά μια, ένα αυτοματοποιημένο μηχάνημα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Μπορεί να κάνει φιλικά και να φέρει σε πέρα σε καθήκοντα ιδιαίτερα περίπλοκα και γρήγορα, αλλά πρέπει να έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις προηγουμένως, έτσι. Λοιπόν, η... αυτά το μηχάνημα το κάνει πάρα πολύ γρήγορα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα καταφέρουν τόσο γρήγορα, ακόμα και αν έχουν εκπαιδευτεί. Τους χρειάζεται χρόνος. Μπορούν να συγκεντρώσουν πάρα πολλά δεδομένα οι μηχανές και τα μηχανήματα, αλλά δεν μπορούν να καταλήξουν γρήγορα σε συμπεράσματα. Είναι δύσκολο να κάνουν, ε, να μαντέψουν, αλλά χωρίς να το κάνω αυτό τυχαία, να μπορούν να συνδυάσουν πραγματικά δεδομένα. Ένα άλλο ζήτημα, το είπε και η Δ. Φέρκερ, θα το πω κι εγώ, είναι θέμα εμπιστοσύνης Πώς ξέρουμε ότι το μηχάνημα θα κάνει πάντα αυτό που θέλετε εσείς να κάνει, αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνη πώς θα χτιστεί. Σίγουρα πολλοί από εσά είσαστε άνθρωποι που μάθατε για την ψηφιακή τεχνολογία. Δεν γεννηθήκαμε με ένα κινητό στην κούνια μας. Εννοείται, είναι πράγματα που τα μάθαμε και αποκτήθηκε αυτή η εμπιστοσύνη με το μηχάνημα που χρησιμοποιούμε. Σιγά σιγά. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Οι παλιοί στρατιωτικοί κοιτούν με επιφύλαξη τέτοιες αυτοματοποιημένε αποφάσεις, γιατί κάποιο διοικητή είναι αυτός ο οποίο πρέπει να πάρει την απόφαση και να είναι σίγουρος ότι ξέρει πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αν ένα μηχάνημα πάρει μια απόφαση, δώσει μια απάντηση, αλλά ο διοικητή δεν μπορεί να ξέρει πώ πήρε αυτή την απόφαση το μηχάνημα, τίθεται θέμα εμπιστοσύνη. Οπότε όταν μιλάμε για την αυτοματοποίηση, είναι ένας προβληματισμός πολύ σημαντικός γιατί πρέπει να είναι δυνατή η επαλήθευση καθόλου τη διαδικασία χρήσης τέτοιων αυτοματοποιημένων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης. Και έχει να κάνει και με πολλά ε, πράγματα που κάνουμε και δοκιμές. Υπάρχουν νέες μέθοδοι που αναπτύσσονται συνεχώ και πρέπει να αναπτυχθούν και άλλες που θα επαληθεύουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις από τα μηχανήματα. Τέλος. Η συζήτηση για τα αυτόνομα οπλικά συστήματα πρέπει να τεθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο γιατί υπάρχουν οι νόμοι της ε, ένοπλης σύγκρουσης που είναι η στρατιωτική στόχη, η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα, οι παράπλευρες επόλειες. Οπότε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες και να ξέρουμε αν τα μηχανήματα μπορούν να τους λάβουν υπόψη τους. Σε κάθε απόφαση που λαμβάνει το ΝΑΤΟ περνάει από έξι διαφορετικά στάδια προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι τηρούμε τους κανόνες και τους νόμους της άνοπλης σύγκρουσης. Οποιοδήποτε αυτόνομο οπλικό σύστημα που συμπεριλαμβάνει μια δυνατότητα απόφασης πρέπει να διασφαλίζει ότι εμπίπτει σε αυτά τα πλαίσια και ακολουθεί τους νόμους ένοπλης σύγκρουσης όπως τους χρησιμοποιούν ή οι στρατηγοί οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα σύστημα είτε είναι απόλυτα αυτοματοποιημένο είτε το χειρίζεται άνθρωπος οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανθρώπους καθ' όλη τη διαδικασία ανάλογα με το πεδίο αρμοδιότητας, ανάλογα με το στόχο και μετά λαμβάνεται η απόφαση ποιο είναι το κατάλληλο σύστημα να φέρει σε πέρα αυτή την, αποφάση, αυτή την απόφαση. Τέτοια μηχανήματα λοιπόν θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές τις προδιαγραφές. Είπα ότι θέλω να είμαι σύντομο, οπότε θα σταματήσω εδώ. Σα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και ελπίζω να σας βοήθησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάλεντα. Συναδελφοί, πρέπει να σας ενημερώσω για τα διαδικαστικά τώρα. Υποχρεωμάστε να τερματίσουμε τη συνεδρίες στις 12.30 ακριβώς. Τουλάχιστον εκεί θα φύγουν οι διερμηνείς. Ε, ε, αλλιώς θα πρέπει να μιλήσουμε αγγλικά αν φύγουν χωρίς ερμηνεία. Δίνω το λόγο στα μέλη που επιθυμούν να μιλήσουν και προτείνω μετά να δώσουμε το λόγο εδώ στον εκπρόσωπο της ΕΕΣ τον κύριο Σύμβουλο και ειδικό απεσταλμένο για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό κυρία Λόζινγκ χωρίς άλλη καθυστέρηση Σας ευχαριστώ πολύ θα μιλήσω γερμανικά, οπότε φορέστε ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, η κυρία Φράνκε, νομίζω πως καταφέρατε να μας ε, δώσετε μία εικόνα της κατάστασης βήμα προς βήμα και να μας φέρετε ε, σε θέση να κατανοήσουμε αυτό το πολύ δύσκολο και πολύπλοκο θέμα και να κατανοήσουμε φυσικά την πολυπλοκότητα του θέματος αυτού. Πρέπει να πω ότι καταφέρατε επίσης να μας δείξετε και τα όρια της επιστήμης και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων πράξεων και της ε, τεχνολογίας. Ε, καταφέρατε να μας δείξετε πράγματα τα οποία εμείς οι πολιτικοί προσπαθούμε ε, να δείξουμε, τις συνέπειες των πράξεών μας δηλαδή. Ε, είχαμε τη, τη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για ε, την κοινή πρόταση ψηφίσματος ε, και θα επικεντρωθούμε στον θανατηφόρο χαρακτήρα των οπλικών αυτών συστημάτων. Και θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως είπατε κι εσείς, να παρουσιάσουμε την αλήθεια, ότι από τη μία τα συστήματα αυτά μπορεί και να κάνουν λάθη, ε, παράλογα λάθη και από την άλλη να ε, αναφέρουμε και ότι τα λάθη αυτά μπορούν να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές και τα λάθη τα οποία προέρχονται από τους ανθρώπους έτσι και αλλιώς. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό και σας ευχαριστώ πολύ που καταφέρατε να το ε, δείξετε. Επίσης, ε, νομίζω πως ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την προκατάληψη, ότι υπάρχουν προκαταλήψεις για αυτά τα ε, συστήματα, τα οποία μάλιστα στην περίπτωση αυτή που μας είπατε από τις Ηνωμένε Πολιτείες ενήργησαν ρατσιστικά θα λέγαμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε και αυτή την πλευρά και το πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον η τεχνητή αυτή νοημοσύνη. Πολύ σημαντική είναι επίσης και η ταχύτητα ε, σε θέματα εξοπλισμού. Γι' αυτό λοιπόν προκύπτει το ερώτημα της ε, ταχύτητας και εάν αυτή η ταχύτητα στον εξοπλισμό θα περάσει και σε άλλους τομείς, ε, αν μπορούν να γίνουν λάθη τα οποία θα λειτουργήσουν καταλητικά για την ε, έκρηξη παγκοσμίου πολέμου. Αυτά ως προς την τεχνική επιτυχή. Θα ήθελα τέλος να επικεντρωθώ στη, στα νομικά ζητήματα, τα οποία εμείς ως πολιτικοί ε, είναι καθήκον μας να αναφέρουμε. Μας είπατε πως ε, ε, υπάρχουν θέματα αποδοτικότητα ε, πως υπάρχουν περιπτώσεις ε, θανάτωσης ε, ανθρώπων. Ακούσαμε και από συνάδελφο για, την, για τις προσπάθειες που γίνονται για την κατάργηση της ε, θανατικής ποινή. Αυτό όμως αντιτίθεται στο ίδιο, στην ίδια τη λογική των οπλικών συστημάτων. Δηλαδή καταδικάζουν σε θάνατο ανθρώπους χωρίς δίκη. Και μα είπατε κι εσείς ότι ο άνθρωπος μπορεί να διστάσει να πατήσει τη σκανδάλη. Τα συστήματα αυτά όμως όχι. Και αυτές είναι οι συνέπειες ε, που πρέπει να αναλογιστούμε και αυτό συνηγορεί και υπέρ της ε, παγκόσμια απαγόρευσης των ε, αυτών οπλικών συστημάτων. Επίσης, ο κ. σκέλα μα είπε για ε, νόμους σε περίοδο πολέμου ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε κήρυξαν πόλεμο επικαλούμενες τρομοκρατία και ε, κάτω από τον ε, πολεμικό αυτό νόμο ε, το να σκοτώσεις κάποιον επιτρέπεται. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να τα, να τα πούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Γκόμες, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φράνκη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επισκόπηση και πολύ κρίσιμα τα ερωτήματα που μας θέτετε. Τίθενται φυσικά νομικά ερωτηματικά, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι το ηθικό που αναφέρατε στο τέλος. Και ήθελα να πω από αυτή την άποψη ότι πολλοί από εμάς προετοιμάζουμε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ελπίζουμε να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα για τα συστήματα αυτά. Τι θα θέλατε εσείς, ε, τι θέση προτείνατε να υπάρχει μέσα σε αυτό το ψήφισμα βάσει των όσων επισημάνατε εδώ. Κατά την απόψη μου προφανώς το κεντρικό ερώτημα είναι μάλλον πρέπει να τα απαγορεύσουμε. Απαγορέψτε τα διεθνώς ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-μέλη και αν χαίρομαι για τις προσπάθειες που έκανε ο κ. Καλέντερ να μας εξηγήσει ότι τα συστήματα αυτά που υπάρχουν δεν ε, είναι τέτοια συστήματα και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις εξελίξεις διότι αποτελούν πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο. Αλλά αν το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ ε, σκοπεύει να εκπληρώσει τους στόχους του, θα πρέπει αμέσως να ξεκινήσει μια εκστρατεία απαγόρευσης των συστημάτων αυτών. Διότι δεν είναι το θέμα του Ηνωμένο Βασίλειο και η πρόληψη δράσεων. Και να λέμε οι ανθρωπιστικές νομοθεσίες είναι αρκετές. Λέτε ότι οι κανόνες για τις ένοπλες σειράξεις και οι σχετικές νομοθεσίες αρκούν. Αλλά αυτά τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εκτός σειράξεων. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πόλεμος. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τρομοκρατικές ομάδες, από οποιαδήποτε ομάδα κακών ανθρώπων, χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο. Έτσι λοιπόν, ε, ξέρετε, ε, οι συνέπειες μπορεί να είναι τρομακτικές. Χαίρομαι που επιβίωσα τον Στανισλάβ Πέτροφ, ο οποίος το 1983 ε, πρόλαβε μια πυρηνική επίθεση χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι δεν αντέδρασε στους συναγερμούς που του έλεγαν ότι επεκτο, επεκτο, ε, ε, τους πλήξει πύραυλος αμερικανικός. Οπότε προτιμώ τον άνθρωπο ως κριτή και όχι το μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα. Και όπως είπατε, το μηχάνημα μπορεί να κάνει λάθη χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη, χωρίς να μπορούμε να το αποδώσουμε ευθύνη. Όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουν σοβαρές προσπάθειες για την απαγόρευση. Γιατί αναπτύσσουν τέτοια συστήματα. Δεν είναι μόνο αμυντική η προσέγγιση, εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Θα ήθελα να το σχολιάσετε κύριε Κάλεντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φρόντ. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομο. Ναι, εν συντομία. Και πάλι σας ευχαριστώ. Πολύ διαφωτιστική συζήτηση που κάναμε εδώ. Επιβεβαιώνει ε, το παλιό ρητό ότι κάθε μέρα μαθαίνει κανείς κάτι καινούριο. Ο κύριος Κάλεντερ και ελπίζω να μην είμαι ο μόνος που το παρατήρησε. Ο κύριος Καλέντερ λοιπόν πολύ έξυπνα περιέγραψε εκτενώς τα όσα δεν έχει το ΝΑΤΟ. Δεν έχει, το τονίζω. Και έτσι μάθαμε πολλά από, αυτές, από αυτά που μας περιέγραψε. Αλλά ήθελα να επιστρέψω στην δόκτωρα Φράγκα και να σας ρωτήσω Πόσο έχει προχωρήσει η ανάπτυξη των όπλων που περιγράψατε. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε, σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα. Ξέρετε, σχεδόν καθημερινά διαβάζουμε για αυτόνομα αυτοκίνητα. Τι μπορεί να επιτευχθεί εκεί, τι σφάλματα υπάρχουν. Μερικές φορές κάνα τέτοιο αυτόνομα αυτοκίνητο σκοτώνει και καμιά ποδηλάτησα. Αλλά αυτό που περιγράφεται για τα όπλα φυσικά είναι πολύ πιο τρομακτικό. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πού βρισκόμαστε σήμερα και αν... Ε, τώρα αυτό σχετίζεται μετά όσα είπαν οι συνάδελφοί μου κυρία και η κυρία Λύση. Μπορούμε να το σταματήσουμε, μπορούμε να προλάβουμε περαιτέρω εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάτσεκ Μπελίτσα σας παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας συγχαίρω και για το θέμα που επιλέξατε. Είναι πραγματικά επίκαιρο όσον αφορά τη στρατιωτική τεχνολογία. Ε, εχμής μάλιστα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις ε, και τον κατάλογο των προβλημάτων που παρέτησε η Δόκτωρ Φρανκ. Εγώ θα προσέθετα και τον κίνδυνο χαμηλώματος του κατοφλίου ε, προσφυγή σε στρατιωτικές ε, παρεμβάσεις και τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας σύρρηξης, διότι τέτοια συστήματα, αν είναι μη επανδρομένα, μειώνουν ε, τον κίνδυνο των απώλειας ανθρώπινων ζώων. Αυτό είναι ο κίνδυνος λοιπόν. Αλλά γίνεται συζήτηση, όπως θέλω να επισημάνω, σε πολυμερή φόρα στο πλαίσιο της σύμβασης για κάποια συμβατικά όπλα στη Γενέβη και υπάρχει μια ομάδα κρατικών εκπροσώπων που τα συζητούν αυτά και οι κυβερνήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούν έτσι να καταλήξουν σε κάποια στοιχεία κοινή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ευρωπαϊκέ θέσει ε, των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι πρέπει να γίνει από αυτή την άποψη. Ειδικότερα, εμεί το επικυρώνουμε, αποτελεί κεντρικό στοιχείο τη ε, θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το, το με αυτόν. Επικοινωνούμε λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και έτσι τονίζουμε τη σπουδαιότητα, τη σημασία του ελέγχου από ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφασίζουν κατά πώς θα χρησιμοποιηθούν θανατηφόρα όπλα. Οι άνθρωποι θα πρέπει να ελέγχουν αυτά τα θανατηφόρα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν και αυτοί θα πρέπει να διατηρούν την ευθύνη αποφάσεων ε, Ζωή λοιπόν, η θανατου ο σωστό λοιπον ανθρώπινο έλεγχο ειναι σημαντικότατο ωστε να διασφαλιζεται η συμμορφωση με τι ε, θεμελιώδει αρχέ ε, του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, θα ήθελα να επισημάνω μια άλλη διαδικασία που ήδη τρέχει σε πολλά από τα κράτη-μέλη μα. Η διαδικασία του άρθρου 36, όπω ονομάζεται, αναφέρεται στο επιπλέον πρωτόκολλο 1 στο πρόσθετο πρωτόκολλο 1 ε, της ε, Σύμβασης της Γενέβης εφαρμόζεται στο γεγονός ότι νέα οπλικά συστήματα τα οποία αναπτύσσουν τα κράτη-μέλη μας πρέπει να έχουν υποστεί κάποια αξιολόγηση συμμόρφωσης με το διεθνές ε, ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμεί υποστηρίζουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία του άρθρου 36 και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση Και το τελευταίο σημείο που σχετίζεται με την απαγόρευση δεν υπάρχει συμφωνημένη ευρωπαϊκή θέση. Ωστόσο υπάρχει μια πρόταση που υποστηρίζεται τουλάχιστον από ένα από τα κράτη-μέλη μα για μια νομική δεσμευτική απαγόρευση. Βρίσκεται επιτάπητο στη Γενέβη αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη μας προτιμούν κάποιο είδους πολιτική δήλωση, κάποιον ε, κώδικα διοντολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρέσβη. Να δώσω τώρα το λόγο στα μέλη του πάνελ με την ίδια σειρά όπως προηγουμένως. Thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Όλους για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Θα ξεκινήσω από τέλος. Συμφωνώ ότι τα θανατηφόρα αυτόνομα ε, όπλα αλλάζουν τα δεδομένα της ε, εμπόλεμη σύραξης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να κάνουμε έρευνες και να δούμε κατά πόσο ευσταθεί αυτό που λέτε, όμως ε, γνωρίζω ότι πράγματι ε, είναι δυνατόν και έχετε πάρα πολύ ε, δίκιο για την κλιμάκωση της κατάστασης ακούσια. Υπάρχει λοιπόν όντως κίνδυνος ακούσιας κλιμάκωσης με τη χρήση αυτών των οπλικών συστημάτων. Η κυρία Γκόμες ρώτησε για ε, τον λόγο για τον οποίο αναπτύσσουμε τέτοια συστήματα. Στην παρουσίασή μου αναφέρθηκα σε αυτό. Υπάρχει μια λογική πίσω από αυτή την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων στρατιωτικά, διότι τα συστήματα αυτά αναπτύσσονται διότι είναι πιο γρήγορα, δεν εντοπίζονται, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς ε, χρησιμοποιώντας τα χωρί, ε, που δεν μπορεί να κάνει με ανθρώπους, σας ανέφερα τα σμήνη, ε, drones, άλλες στρατιωτικές ικανότητες που γίνονται δυνατές χρησιμοποιώντας αυτονομία και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό λοιπόν είναι το σκεπτικό πίσω από την χρήση και ανάπτυξή τους και φυσικά, όπως είπα και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από τις λέξεις, ε, της φράσεις κλειδιά της εποχής μας. Ε, όχι μόνο ε, στον στρατό. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται παντού, σε όλους τους τομείς, σε, σε, για πολιτικούς σκοπούς και μετά... Δεν αποκλεί κανείς ότι αυτή η πολιτική τους χρήση θα έχει στρατιωτικά ωφέλη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να περιορίσουμε τη χρήση τους, ακριβώς για αυτήν την διπλή χρήση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση, κατανοώ το σκεπτικό πίσω από, τους, ε, από τις οργανώσεις και τις ομάδες που ζητούν απαγόρευση των αυτόμα, αυτόνομων συστημάτων, όμως ε, ε, επιτρέψτε μου κάποιες αμφιβολίες. Καταρχάς, υπάρχει το πρόβλημα της διπλής χρήσης. Δεν πρόκειται και ούτε θα έπρεπε να εμποδίσουμε την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ε, θα ήταν όμως ε, πολύ εύκολο να γίνει διπλή χρήση και είναι δύσκολος ο διαχωρισμός να μην χρησιμοποιείται δηλαδή για στρατιωτικούς σκοπούς ε, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για πολιτικούς. Φυσικά και αναφέρομαι στις, ε, στην περίπτωση τρομοκρατικών οργανώσεων που δεν πρόκειται να φοβηθούν από την απαγόρευση. Η απαγόρευση ζητείται ακριβώς ε, διότι κάποια συστήματα που χρησιμοποιούνται τώρα θα ε, στην απαγόρευση αν εφαρμόζονταν αυτή η νομοθεσία και όσο προχωράμε στο φάσμα προς την πλήρη αυτονομία θα ε, πρέπει να έχουμε επίγνωση του ότι αν απαγορεύσουμε ένα, δεν θα, ένα σύστημα δεν θα απαγορεύσουμε τη χρήση γενικότερα των, ε, της τεχνητής νοημοσύνης και των αυτόνομων συστημάτων. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις συστάσεις, να εστιάζουμε σε αυτά που μπορούμε ή όχι να χρησιμοποιήσουμε και όχι στην εξέλιξη τεχνολογίας καθ' αυτή. Δύσκολο βέβαια, διότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει ότι στόχο έχει τη διασφάλιση επαρκούς ανθρώπινου ελέγχου σε συστήματα που έχουν κάποιο βαθμό αυτονομία στη λειτουργία τους. Και όπως σας είπα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Ε, πράγμα, αλλά χρειάζεται ανθρώπινη υποπτία και έλεγχο. Και προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση, να γίνει δημόσια διαβούλευση ε, για ε, γενικότερα την τεχνητή νοημοσύνη. Νωρίτερα επίσης αναφέρθηκε το ζήτημα εμπιστοσύνης. Μπορούμε να εμπιστευτούμε έναν υπολογιστή αν χρησιμοποιεί τεχνητή νομοσύνη Στην ουσία τι συμβαίνει. Οι υπολογιστέ δεν κάνουν λάθη. 2 και 2 ίσον τέσσερα. Μπορούμε να του εμπιστευτούμε 100%. Όμω τη στιγμή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη αυτό πάβει να ισχύει. Επαναλαμβάνω, τα συστήματα αυτά είναι εξαιρετικά ευφυή, ευφιέστερα από του ανθρώπου, όμω μπορεί να είναι προκατελημένα και να κάνουν λάθη. Γι' αυτό προτείνω η κοινωνία στο σύνολό τη να προσεγγίσει το θέμα αυτό διαφορετικά και να το αντιμετωπίσει όπως το αντιμετωπίζουν, όπως ας πούμε θεωρούμε πως είναι ένας εμπειρογνώμονας. Κάποιος δηλαδή που ναι μεν ξέρει πολύ περισσότερο από μένα για αυτό το θέμα, χωρίς όμως να πάψει να το αμφισβητεί. Ναι λοιπόν, αλλά να κάνουμε και ερωτήσεις. Τώρα, ρωτήθηκα για την πρόοδο της τεχνολογίας. Πού είμαστε. Πολλά μπορούν να γίνουν, πολλά είναι δυνατά, έχουν ήδη γίνει έρευνες, εργαστήρια και δοκιμές εξωτερικές. Μπορούμε να δούμε και στο YouTube, για παράδειγμα, τεράστια σμήνη τέτοιων ε, drones μαχητικών ε, μη επανδρομένων σκαφών στην Αυστραλία ε, που χτυπούσαν στόχους, τους εντόπιζαν. Τα συστήματα αυτά ήδη χρησιμοποιούνται και έχουν δοκιμαστεί. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας, εξαρτάται ε, τι θεωρείτε αυτόνομο ε, σύστημα. Το σύστημα Harpy του Ισραήλ είναι ας πούμε μια τέτοια περίπτωση. Ε, που εντοπίζει στόχους και ραντάρ. Το Αζερβαϊτζάν επίσης, παρεπιπτόντος, χρησιμοποίησε το σύστημα αυτό όχι όμως για να εντοπίσει ραντάρ, αλλά το χρησιμοποίησε εναντίον ενός λεωφορείου ε, γεμάτου με ε, ε, στρατιώτες από την Αρμενία. Όπως βλέπετε λοιπόν, μπορείμε να μην έχουμε φτάσει σε επίπεδα εξολοθρευτή, όμως βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να προχωράμε προς την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα οπλικά συστήματα, στη χρήση αυτόνομων συστημάτων. Γι' αυτό λοιπόν και νομίζω πως η ερώτηση πρέπει να είναι για τα όρια, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Πού σταματάμε, θα ε, σταματήσουμε πριν πάρουμε την απόφαση να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κάλαντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. δεν έχω πολλά σχόλια, διότι δεν ε, ε, είμαι σε θέση, δεν είναι ο μου να εκφέρω απόψεις. Ε, τώρα, όταν μιλάμε για τις ευρωπαϊκές χώρες που ασχολούνται με την τεχνητή νομοθεσία, Πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν και η τεχνητή νοημοσύνη ορίζει τι μπορούμε να κάνουμε για τα συστήματα αυτά από υπολογιστική άποψη, αλλά με αυτό σχετίζεται και η αυτονομία. Ποιες πλατφόρμες ε, ε, τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνονται για να γίνει οτιδήποτε. Ε, μιλάμε για ένα τεράστιο φάσμα στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ρομποτικά συστήματα που φτιάχνουν αυτοκίνητα, ε, μέχρι μη επανδρομένα ε, αεροσκάφη, ε, υπτάμενα αντικείμενα που κινηματογραφούν ας πούμε παρελάσεις, αγροτικές τεχνικές, αγροτικά συστήματα και στρατιωτικές εφαρμογές. Η εφαρμογή λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανικά και εμπορικά συστήματα είναι ευρεία. Αλλά δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τι κάνουν τα κράτη-μέλη το καθένα όσον αφορά τα αυτόνομα οπλικά συστήματα. Αλλά η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει στα περισσότερα κράτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ και τα μέλη του Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο Μπελίτσα. Ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα παρουσιάσουμε ένα ψήφισμα επιτέλους το οποίο διαπραγματευτήκαμε ήδη το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες ε, ε, ένα ψήφισμα για τα ΛΟΟΖ θα γίνει και ψηφοφορία λοιπόν και στην επόμενη σύνοδό μας τον Οκτώβριο από όσο θυμάμαι στις 10 Οκτωβρίου θα έχουμε μία ακρόαση εντός της ΕΝΤΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε παρακαλώ να είστε παρόντες. Τα... Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν τους ομιλητές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία, τους δερμηνείς και να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ.